Καλησπέρα σα. Αγαπητοί συνάδελφοι. Σαν αρχίζω το σχολείο, αισθάνομαι. Πρώτη μέρα στο σχολείο. Καλησπέρα σας. Αν δεν έχετε σχόλια, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Καταρχά, σα καλωσορίζω στην πρώτη αυτή συνεδρία τη ΕΜΗΣ. Είμαι πεπισμένη ότι πρόκειται αυτή η χρονιά να αποδεχθεί πολύ επικοδομητική, με ενδιαφέρουσε και εντατικέ ακρόασει για όλους μας. Καλά αποτελέσματα και μια πολύ καλή έκθεση για να κλείσουν οι εργασίε. Ξέρετε ότι έπρεπε να έχει γίνει η πρώτη μα ακρόαση στι 22 Μαρτίου, λόγω όμω των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα τη μέρα εκείνη στις Βρυξέλλες χρειάστηκε να ματαιωθεί. Φαντάζομαι να το να αντιλαμβάνεστε και να δείχνετε κατανόηση. Εγώ προσωπικώς δεν θα μπορούσα να πω ούτε μια κουβέντα με ηρεμία εκείνη τη μέρα. Ελπίζω βέβαια αυτή η καθυστέρηση να μην οδηγήσει σε οποιαδήποτε ε, περίπλοκη των εργασιών της ε, Επιτροπής μας. Έχουμε 15 γλώσσες στη διερμηνία. Έχουμε μετάδοση μέσα από το διαδίκτυο και το Europal TV και το ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο πνεύμα της των λιγότερο χαρτιού τα έγγραφα τα έχετε σε σας ηλεκτρονικά πρακτικά της 10ης και 16ης Μαρτίου συνεδριάσεων συντονισμού. Είναι στη θέσή σας. Έχει δημοσιευθεί, θα δημοσιευθεί και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στην ιστοσελίδα, ε, στον ιστότοπα μας προκειμένου να έχουμε ε, να το μεγαλύτερη διαφάνεια. Ξέρετε ότι είναι δύσκολο να βρούμε χρόνο με δεδομένη την ε, δουλειά την ίδια εβδομάδα που συνεδριάζουν και άλλες επιτροπές. Είναι δύσκολο να βρεθεί ο χρόνος για τη δική μας επιτροπή. Θα δείτε καμιά φορά συνεδρίαση πέμπτη απόγευμα, αναγκαστικά. Σας παρακαλώ να δείξετε και σε ευελιξία και να προσαρμόσετε ανάλογα το πρόγραμμα των εργασιών σας. Θα είναι πολύ εντατική η φετινή χρονιά. Οι συστατικοί συνεδρίες με τα πρακτικά της σας έχουν κατατεθεί. Πρόκειται για την συνεδρίαση Δευτέρα Μαρτίου, αν δεν έχετε αντίρρηση εγκρίνονται και, ε, αν δεν έχετε αντίρρηση, περνώ στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης που αφορά την ανταλλαγή. Παρακαλώ. Κυρία Βάλτερ Μόζα, μία παρατηρήση. Δεν έχω διερμηνία στα δανέζικα σήμερα. Ελπίζω να μην επαναληφθεί αυτό στο μέλλον, γιατί χρειάζομαι τη διερμηνία. Η Πρόεδρος. Ναι, Ολλανδικά, Ολλανδικά. We'll take that with us. Um, το σημειώνουμε. αλλά εξαρτάται και από το γεγονός ότι ήμασταν ε, η τελευταία ε, συνεδρίαση που εγγράφηκε στο πρόγραμμα των Επιτροπών. Και η αίθουσα μας δεν είναι από τις πιο μεγάλες υπάρχουν διάφορε ποσοστώσει και τα λοιπά από ό,τι μαθαίνω. Το σημειώνουμε πάντως, για να μπορεί να κάνει ο καθένα τη δουλειά του σωστά. Και πάω στο σημείο 4. Ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη, Γενική ε, Διεύθυνση για την ε, Κλιματική Αλλαγή και για το περιβάλλον. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι προσεχείς συνεδριάσεις θα δουν και την πρόσκληση μαρτύρων, όπως απαιτείται κανονικά σε μια εξεταστική επιτροπή. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Σήμερα έχουμε την παραδοσιακή τυπολογία της ακρόασης, δηλαδή μια ανταλλαγή περισσότερων απόψεων με εκπροσώπους των ε, Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής σήμερα. Ενδέχεται όμως τους ίδιους ή άλλους να τους δούμε υπό την ιδιότητά τους ως εργαζομένων σε αυτό ή τον άλλον τομέα και ως μάρτυρες κάποια στιγμή. Αυτό είναι τώρα για να ξεκινήσουμε, για να είμαστε ενήμεροι όλοι από την ίδια βάση και να ξεκινήσουμε όλοι με ισότιμες ε, δυνατότητες αυτή τη δουλειά. Έχουμε περίπου δύο ώρες προβλέψει δεν ε, με χαρακτηρίζει αυτό, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι στο δυνατόν πιο προσεκτική ως προς το χρόνο ως πρόεδρος, γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τη σημερινή συνεδρία, αλλά ιδιαίτερα για τις ακροάσεις με τους μάρτυρες. Εκεί θα χρειάζεται να τηρούσουμε με αυστηρότητα το χρόνο περισσότερο. Καλώς ορίζω λοιπόν τον πρώτο μιλητή. Θα ακούσουμε πρώτα τους ομιλητές, πρέπει να θα έρθουν οι ερωτήσεις. Ο κύριος Αντίπελ Τομάκη, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ιστορικής Αγοράς, Βιομηχανίας Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, της Γενικής Διεύθυνσης για την Ανάπτυξη δηλαδή, της GROW. Θα μας μιλήσει για το σύστημα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος έγκρισης της ε, τυπολογίας και θα διευκρινίσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών στην τήρηση των προδιαγραφών των σχετικών με τις εκπομπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Αντιπρόεδροι, αξιότιμα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πω ότι είμαι ικανοποιημένο και ευχαριστημένο που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα, αλλά τουλάχιστον Είμαι σε θέση να σας πω ότι μπορώ πλέον να συμβάλλω σε εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής που ξεκινάει σήμερα τις εργασίες της και όπως είπατε κι εσείς κυρία Πρόεδρε, προσπαθώ να καλύψω διάφορα ζητήματα τα οποία αναφέρατε κι εσείς ε, στην εισαγωγική σας παρέμβαση. Ήδη από το 2007, από τότε που εγκρίθηκαν οι κανονισμοί γύρω 5 και γύρω 6, πολλά πράγματα έχουν γίνει και φτάσαμε σήμερα στον, στη δικασία δοκιμής RDE, Real Driving Emission, εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Για ποιο λόγο επιλέξαμε αυτή την προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Ήδη θα ήθελα να σας πω ότι θεωρήσαμε ότι αυτή ήταν η καλύτερη προσέγγιση προκειμένου να έχουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε απόπειρα εξαπάτηση στο σύστημα εκπομπών. Το σύστημα αυτό επίσης, το RDE, δεν θα πρέπει να το δούμε απομονωμένα. Αποτελεί τμήμα της γενικότερης δέσμης μέτρων μαζί με τη μεταρρύθμιση του συστήματος έγκρισης τύπου και πιστεύουμε ότι αυτή η νέα δέσμη μέτρων θα μας δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα και αυτό περιμένουν άλλωστε και Ευρωπαίοι πολίτες. Θα ήθελα επίσης στη συνέχεια να καλύψω και τον όλο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τις εκπομπές και ιδίω την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κρίση Volkswagen. Και προκειμένου να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ποιο είναι ο ρόλο τόσο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και των κρατών μελών, θα πρέπει να βρεθούμε περισσότερο σε ζητήματα εφαρμογή τη νομοθεσία μα. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ορισμένα πράγματα όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο για την έγκριση τύπου συστήματος, πώς έχει αυτό δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Όπω ξέρετε, το σύστημα αυτό είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι εθνικέ αρχέ πιστοποιούν ένα μοντέλο αυτοκινήτου προτού αυτό διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και λένε ουσιαστικά ότι συμμορφώνεται με όλε τι περιβαλλοντικέ απαιτήσει και τι απαιτήσει ασφάλεια. Επικεντρώνεται σε συγκεκριμένου έλεγχου που γίνονται πριν διατεθεί το προϊόν αυτό στην αγορά ήδη από την φάση κατασκευής του και στην αρμολόγησή του στο εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή εγκριθεί σε ένα κράτος μέλος μπορεί να διατεθεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν ένα κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά από την άλλη οι εθνικές αρχές οφείλουν και αυτές να ελέγχουν την συμμόρφωση των κατασκευαστών αυτοκινήτων και για το ζήτημα των εκπομπών. Κάποιες τώρα ρηπογόνες ουσίες, όπως για παράδειγμα τα οξύδια αζότου, οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα ανήκουν πλέον σε ένα σύστημα το οποίο το ονομάζουμε NEDC. Εκεί πέρα ελέγχονται. Πρόκειται για ένα νέο κύκλο δοκιμών όσον αφορά τι εκπομπέ κατά τη διάρκεια τη οδήγηση. Ήδη από το 1990 έχει σχεδιαστεί το σύστημα αυτό και ουσιαστικά αναφέρεται σε κάποιε νέε μορφέ επιτάχυνση που εμφανίζονταν στα αυτοκίνητα. Βλέπουμε όμως ότι οι έλεγχοι αυτοί που γινόντουσαν αποκλειστικά σε εργαστήριο είναι αρκετά περιορισμένοι και δεν ανταποκρίνονται πάντα σε αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Υπήρξε ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο χάσμα ανάμεσα στι πραγματικέ εκπομπέ και τι εκπομπέ τι οποίε μπορούσαμε να μετρήσουμε στα πλαίσια του εργαστηρίου, ιδίω όσον αφορά το οξύδιο του αζότου και το διοξίδιο του άνθρακα. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία δοκιμών, προκειμένου να έχουμε πιο ακριβείς μετρήσεις των εκπομπών και κατά αυτόν τον τρόπο να ανταποκρινόμαστε περισσότερο στην πραγματική κατάσταση εργαζόμαστε σε δύο πτυχές. Από τη μία πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, στα πλαίσια του UNEC συγκεκριμένα, προκειμένου να δημιουργηθεί το WLTP, δηλαδή μια νέα παγκόσμια διαδικασία δοκιμής των εκπομπών στα ελαφρά οχήματα και θεωρούμε ότι με το νέο αυτό σύστημα θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τι μετρήσει που γίνονται για τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Και από την άλλη κάνουμε κάποιε περαιτέρω δοκιμέ προκειμένου να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο θα επιτρέπει να κάνουμε ακριβεί μετρήσει όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα και τα οξύδια του αζότου σε πραγματικέ συνθήκε οδήγηση. Θα ήθελα τώρα να περάσω στην διαδικασία RDE, εκπομπέ σε πραγματικέ συνθήκε οδήγηση και τι σχετικέ δοκιμέ. Από τότε που εγκρίθηκε ο κανονισμός γύρω 5 και γύρω 6, από το 2007 δηλαδή, άρχισε να εφαρμόζεται σε νέες μορφές οχημάτων του τύπου Euro 5 ήδη από το Σεπτέμβριο του 2009. Φάνηκε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τότε είχε συνειδητοποιήσει ότι η μέτρηση των εκπομπών στο εργαστήριο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική μέτρηση των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί μια νέα νομοθεσία που θα μας επιτρέπει να κάνουμε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτό το νέο σύστημα RDE βάσει μελετών και ερευνών που γίνανε από διάφορα ερευνητικά κέντρα αλλά και από το JRC, το Εσωτερικό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, πολλοί εμπειρογνώμονες συμμετείχαν στην Τεχνική Επιτροπή για τα μηχανοκίνητα οχήματα TCMV, η οποία μετά από 3,5 χρόνια κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Χρειάστηκε επίσης ένας ακόμα χρόνος προκειμένου τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της Τεχνικής Επιτροπής για τα μηχανοκίνητα οχήματα να καταφέρουν από πολιτικής πλευράς πλέον να μια συγκεκριμένη πρόταση. Κάθε φορά που γίνονται συζητήσεις για το ζήτημα αυτό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφερόμαστε και στην παραληφθούσα συμμετοχή του Κοινοβουλίου, το οποίο μπορούσε να ελέγχει όλες αυτές τις διαδικασίες και ήδη από το 2016 έχει μεγαλύτερο ρόλο στον έλεγχο των νέων αυτών συστημάτων που χρησιμοποιούνται. Πώς θα λειτουργήσει το νέο αυτό σύστημα θα χρησιμοποιηθούν φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών, τα οποία θα είναι σωματωμένα στα οχήματα και κατά αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί πάρα πολύ το χάσμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις πραγματικές εκπομπές και τις εκπομπές όπως αυτές εμφανίζονται στο εργαστήριο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί και οποιαδήποτε δυνατότητα χρησιμοποίησης συσκευών εξαπάτησης, defeat devices. Κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιληφθεί πλήρως του ζητήματος αυτού. Για ποιο λόγο ακολούθησε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προσέγγιση αυτή. Ήδη στου κανονισμούς γύρω 5 και γύρω 6 είχαμε διάφορες εξουσίες που μας δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε τις επιμέρους αυτές διατάξεις που υπήρχαν στους κανονισμούς αυτούς. Προβλεπόταν επίσης και η δυνατότητα δημιουργία νέων δοκιμών για τα συστήματα έγκριση τύπου, καθώ επίση και για την ε, αναθεώρηση του συστήματο μέτρηση εκπομπών. Εξ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να καταλήξει συγκεκριμένα συστήματα μέτρησης προκειμένου να μην είναι δυνατή χρησιμοποίηση οποιασδήποτε συσκευή εξαπάτησης. Από τεχνικής πλευράς αυτό ήταν δύσκολο και αυτό φάνηκε και από τις μελέτες του JRC. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εστιαστεί περισσότερο στην ανάπτυξη ενός ισχυρού συστήματος RDE γιατί θεωρήθηκε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα διασφάλιζε από τη μία πλευρά ότι θα έχουμε όντως ε, δοκιμές ε, εκπομπών οι οποίε θα ανταποκρίνονται στις πραγματικέ συνθήκε οδήγηση και από την άλλη δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε συσκευές εξαπάτησης εύκολα. Σε διαβούλευση με, τους, με τα ενδιαφερόμενα μέρη κάναμε συγκεκριμένες νομοθετικές επιλογές. Ακολουθήσαμε επίσης τις συστάσεις διαφόρων ε, ερευνητικών φόρουμ, όπως για παράδειγμα η Υψηλόβαθμη ομάδα εργασίας CARS 21 και 2020. Και χρησιμοποίησαμε επίσης και τη συμβολή των κρατών μελών της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και κάθε φορά με τις σχετικές εκθέσεις και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεριέλαβε τις παρατηρήσεις αυτές σε ένα ψήφισμά του τον Νοεμβρίου του 2013 συγκεκριμένα δηλαδή με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το, τη δέσμη μέτρων CARS 2020. Πρέπει να είμαι ξεκάθαρο στο σημείο αυτό. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε πλήρες συνθήκες συνένεσης, γι' αυτό προχωρήσαμε και σε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής όμως ότι ε, σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακολουθεί τις απαιτήσει ε, συγκεκριμένων συμβαλωμένων ε, μερών αν δείτε πραγματικά ποιε ήταν οι νομοθετικέ μας επιλογές, ιδίω όσον αφορά το RDE testing, θα δείτε ότι έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από την προτινόμενη επιλογή του συγκεκριμένου κλάδου, του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Για ποιο λόγο τώρα άργησε τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει αυτό το νέο σύστημα δοκιμών, RDE. Είπαμε ότι χρειάστηκαν περίπου 3,5 χρόνια προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη η τεχνική εργασία και επιπλέον ένας χρόνος στη συνέχεια για να ληφθεί μια απόφαση σε πολιτικό επίπεδο. Δεν νομίζω όμω ότι μπορεί κανεί να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση στο τι αποτελεί αποδεκτό χρονοδιάγραμμα. Θεωρήσαμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουμε τον απαραίτητο χρόνο στην επιστημονική έρευνα, να συλλέξουμε και να συγκρίνουμε τεχνικά δεδομένα και να αξιολογήσουμε διαφορετικέ μεθόδου για τη μέτρηση των εκπομπών, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα ισχυρό σύστημα από τεχνική πλευρά. Πέρα όμω από την τεχνική αυτή πλευρά, όπω σα είπα, έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητε διαβουλεύσει με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αν συγκρίνουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα λοιπόν με πρώτερες εμπειρίες που είχαμε όσον αφορά κυρίως τα βαρέα οχήματα, τότε βλέπουμε ότι σε προηγούμενες περιπτώσεις είχαν χρειαστεί περίπου 8 χρόνια. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η διαδικασία RDE είναι μια διαδικασία αρκετά πολύπλοκη που δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε κανένα άλλο νομικό σύστημα παντού, πουθενά στον κόσμο. Η διαδικασία αυτή RDE δοκιμή δηλαδή μέτρηση των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγηση, είναι αν θέλετε μόνο η αρχή της ιστορίας. Προτείνουμε αυτή τη στιγμή τέσσερι διαφορετικέ νομοθετικέ πράξεις όσον αφορά την μέτρηση των εκπομπών. Η δεύτερη νομοθετική αυτή πράξη έχει να κάνει με τις ποσοτικές απαιτήσει για τι εκπομπέ οξυδίου αζότου κατά τη διάρκεια των δοκιμών RDE. Και αυτό γίνεται καθορίζοντας του παράγοντε συμμόρφωση και για να είμαι πιο συγκεκριμένο, είναι αυτοί οι παράγοντε συμμόρφωση οι οποίοι καθορίζουν τα ανώτατα όρια τιμών, αυτά τα οποία ονομάζουμε not to exceed limits, και αυτό σε όλε τι μορφέ RDE testing. Όπω για παράδειγμα, ακόμα και όταν ένα όχημα ανεβαίνει μία ανηφόρα με πολύ μεγάλη κλίση. Καταλήγουμε λοιπόν στις μέσες τιμές οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές σε φυσιολογικές συνθήκες οδήγησης. Η δεύτερη επίση αυτή νομοθετική πράξη RD δημιουργεί συγκεκριμένε υποχρεώσει για του ε, κατασκευαστέ οχημάτων όσον αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν για τη μείωση των εκπομπών. Και κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούν να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε ευελιξία ενδεχομένω είχαν στα πλαίσια των δοκιμών που γινόντουσαν στα εργαστήρια. Η τρίτη τώρα νομοθετική πράξη RD θα έχει ω στόχο την μέτρηση των ρηπογόνων σωματιδίων, ενώ η τέταρτη σχετική νομοθετική πράξη θα ζητά από την αυτοκινητοβιομηχανία να δημοσιοποιούν όλες ε, τις, όλους τους παράγοντες συμμόρφωσης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα διάφορα πιστοποιητικά συμμόρφωσης COC τα οποία ε, δημοσιοποιούν οι διάφορες ε, εταιρείες. Στην περίπτωση της Volkswagen βλέπουμε ότι το Type Approval System που είχαμε στο παρελθόν, το σύστημα έγκρισης τύπου, είχε συγκεκριμένα όρια και περιορισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τις 27 Ιανουαρίου του 2016 έχει προτείνει μια γενική αναθεώρηση όλου του συστήματος έγκρισης τύπου. Σύμφωνα με το παρόν σύστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει απλώς νομοθετικό πλαίσιο, ενώ η εφαρμογή τελικά εναπόκειται εξ ολοκλήρου στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει κανέναν ουσιαστικό έλεγχο όσον αφορά τα οχήματα. Εναπόκειται μόνο στις εθνικές αρχές των κρατών μελών να κάνουν ελέγχους για να δουν αν συμμορφώνονται οι κατασκευαστές αυτοκινήτων και μεταξύ τους μόνο μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τα συστήματα έγκρισης τύπου. Οι περισσότεροι έλεγχοι μάλιστα γίνονται προτού τα οχήματα διατεθούν στην αγορά και πολύ λίγοι έλεγχοι γίνονται όταν τα οχήματα όντως βρίσκονται στην αγορά. Επίσης είναι τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία στα πλαίσια του εθνικού δικαίου καθορίζουν τις ανώτατες ποινέ και τις εφαρμόζουν. Η νέα λοιπόν αυτή πρόταση όσον αφορά τα συστήματα έγκριση τύπου αλλάζει αυτά τα δεδομένα. Προβλέπεται ένα νέο σύστημα το οποίο με μεγαλύτερη διαφάνεια θα εντοπίζει τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες, στις οποίες δεν υπάρχει συμμόρφωση και μάλιστα προτού τα οχήματα διατεθούν στην αγορά. Κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να συμμετέχει άμεσα τόσο πριν όσο και μετά τη διάθεση στην αγορά συγκεκριμένων οχημάτων. Επίσης, προβλέπονται και κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου όλα τα υπεύθυνα, όλοι οι υπεύθυνοι φορεί για την εφαρμογή τη νομοθεσία να λαμβάνουν τι ευθύνε του κατά τρόπον ρομανισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση, θα ενισχυθούν οι φορεί δοκιμών, δεν θα υπάρχουν πλέον εμπορικοί σύνδεσμοί του με του κατασκευαστέ και θα υπάρχει κοινή αξιολόγηση από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, θα υπάρχει ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανακλήσεων οχημάτων σε περίπτωση μη συμμόρφωση, το οποίο θα ισχύει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ε, η ασφάλεια και η υγεία τόσο των καταναλωτών όσο όμως και του περιβάλλοντος θα προστατευτεί καλύτερα. Δημιουργώντα ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τα συστήματα έγκριση τύπου και έχοντα και τα νέα δεδομένα όσον αφορά τις δοκιμές RD, e, δηλαδή τις δοκιμές για τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, δημιουργούμε νέες δεσμεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να αποφεύγουμε παρατυπίες όπως αυτή της Volkswagen. Επίσης θα έχουμε νέες διαδικασίες δοκιμών σε επίπεδο εργαστηρίου αυτή τη φορά, προκειμένου να μετράμε καλύτερα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και τις εκπομπές άλλων τρυπογόνων ουσιών. Κατά αυτόν τον τρόπο θα εναρμονιστούμε καλύτερα και με το σχετικό σύστημα το οποίο υπάρχει σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίσουμε ότι οι εκπομπέ οι οποίε την χάνουν μέτρηση πραγματικά ανταποκρίνονται στι πραγματικέ εκπομπέ σε πραγματικέ συνθήκε οδήγηση. Επίσης, όσον αφορά την περίπτωση της Volkswagen. Για ποιο λόγο το δικό μας σύστημα παρατήρησης και παρακολούθησης δεν κατάφερε να εντοπίσει το πρόβλημα, ενώ εντοπίστηκε το πρόβλημα αυτό από τις αρχές των Πολιτειών. Τόσο στι Πολιτείε, όσο και στις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώ απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση συσκευή εξαπάτηση. Απαγορεύεται αυτό από το δίκαιο τόσο το νοσιακό όσο και από το δίκαιο των Πολιτείων Ποιε είναι όμω οι βασικέ διαφορέ που υπάρχουν στο σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σύστημα των ΗΠΑ. Προφανώ υπάρχουν διάφορε συστηματικέ ε, διαφορέ, αλλά η βασική διαφορά έχει να κάνει με την προσέγγιση μα. Η δική μα ευρωπαϊκή προσέγγιση έχει να κάνει με έγκριση τύπου σε συνθήκε ε, ε, πρώτερο τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε ασχολούνται πάρα πολύ και με το μετέπειτα στάδιο, αφού δηλαδή το όχημα περάσει στην αγορά. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι το σύστημα των ΗΠΑ έχει να κάνει περισσότερο με ουσιαστική παρακολούθηση της αγοράς, και πάλι δεν εντοπίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο για αυτό το λόγο το σκάνδαλο της Volkswagen. Ήταν μη κυβερνητικέ οργανώσεις αυτές οι οποίες κάνανε τις απαραίτητες έρευνες και οι οποίες παρήχανε τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία καταδεικνύανε ότι όντως κάτι δεν πήγαινε καλά με τη Volkswagen και στη συνέχεια βέβαια αυτό προσέγγισε το ενδιαφέρον και των Αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών. Επίσης, στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει ένα ήδη κεντρικό σύστημα προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής της οικολογικής νομοθεσίας, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 28 διαφορετικές αρχές που ασχολούνται με τη συμμόρφωση των οχημάτων. Επίσης, οι περισσότεροι έλεγχοι γίνανε προτού διατεθεί το προϊόν στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπαμε, και πολύ λίγοι έλεγχοι γίνανε μετέπειτα, όταν το, τα αυτοκίνητα πέρασαν στην αγορά, ενώ αντίθετα οι ΗΠΑ ασχολούνταν και με αυτό το στάδιο του ελέγχου. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στιγμή έχει πολύ περιορισμένε δυνατότητε επιβολή του νόμου, ενώ οι ΗΠΑ έχουν στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα νομικά μέσα προκειμένου να επιβάλλουν την νομοθεσία και να απαγορεύσουν συσκευέ εξαπάτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνώριζε ότι οι αρχές εποπτείας σε εθνικό επίπεδο δεν λειτουργούσαν αποτελεσματικά και πλήρως, δεν λειτουργούσαν με ικανοποιητικό τρόπο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο αρχίσαμε ήδη αρκετά νωρί να επενθυμίζουμε στα κράτη-μέλη τι πρέπει να κάνουν. Στείλαμε πάρα πολλές επιστολές στις εθνικές αρχές ήδη από το 2012. Στις επιστολές αυτές ζητούσαμε από τις εθνικές αρχές εποπτείας να εξασφαλίσουν ότι όντω το νέο σύστημα έγκριση τύπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο και ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμένο ε, τρόπο έγκριση τη συμμόρφωση των αυτοκινητοβιομηχανιών. Ακριβώ επειδή υπήρχαν όμω όλε αυτέ οι ελλείψει, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια φιλόδοξη νομοθετική πρόταση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε περισσότερου ελέγχου στα πλαίσια τη αγορά και να κάνουμε περισσότερες συστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανάλογες βελτιώσεις έχουμε κάνει και για το σύστημα έγκρισης τύπου α, τρακτέρ και μηχανών μοτοσακό όπου έχουμε χρησιμοποιήσει περισσότερους πλέον συντονισμένους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μετά το σκάνδαλο της Volkswagen, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη να κάνουν τις απαραίτητες έρευνες και επιθεωρήσεις και να υποβάλουν εκθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκολύνει αυτή την ανταλλαγή στοιχείων ανάμεσα στα κράτη-μέλη και χρησιμοποιεί μια κοινή μεθοδολογία. Μετά τη νέα νομοθεσία για την μέτρηση του διοξιδίου του άνθρακα, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα συγκεκριμένη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη-μέλη να κάνουν ευρύτερε έρευνε για να δούμε αν τυχόν υπάρχουν παραβιάσεις κοινοτικής νομοθεσίας. Βλέπετε ότι όλοι θέλουμε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα και μια απόλυτα διαφανή εικόνα. Επίσης, ξεκινήσαμε διαδικασίες προ... προτού προχωρήσουμε σε επίσημη διαδικασία επί παραβάση απέναντι σε, 23 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όντως εφαρμόζεται σωστά το κοινοτικό σύστημα έγκρισης τύπου. Μπορούμε νομίζω κατά αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε καλύτερα το ρυθμιστικό μας πλαίσιο. Και τέλος, να σας πω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί διατίθεται να δείξει πλήρη διαφάνεια, να συνεργαστεί πλήρω μαζί σα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασκεδαστούν όλε οι ανησυχίε. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν κοινού στόχου όσον αφορά τη διαδικασία αυτή. Επιθυμούμε και οι δύο να βελτιώσουμε το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό σύστημα και θέλουμε το νέο αυτό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό σύστημα να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντο και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον κύριο Καλιέχα. Ελπίζω ότι ε, προφέρω σωστά το όνομά σας από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, τη Γενικός Διευθυντής και θα μας μιλήσετε για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρήμανσης στην ε, ανθρώπινη υγεία. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Είμαι ο Γενικός Διευθυντής ε, της για το περιβάλλον. Οπότε από δική μου πλευρά ε, να σας πω πώς έχει το τοπίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε την πλήρη εικόνα. Και αφετηρία θα έχω το ότι η ρήπανση του αέρα και η επιπτώση στην ανθρώπινη υγεία παραμένει ένα πολύ σημαντικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ε, βασικό πρόβλημα μας απασχολεί. Έχουμε 400.000 πρόωρους θανάτους οι οποίοι προκαλούνται από την ρήπανση του αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο. Και δεν πρόκειται μόνο για αυτούς τους πρόωρους θανάτους. Έχουμε και ένα σωρό ασθένειες, έχουμε απουσιασμό από την εργασία, τέλος πάντων ε, απώλεια παραγωγικότητας και άλλη ζημία και βεβαίω ε, όλα αυτά κοστίζουν πάρα πολύ στο συστήματα υγεία. Η πρωταρχή ευθύνη για την προστασία των ε, πολιτών ε, είναι αρμοδιότητα των εθνικών αργών. Όμως μόνα του δεν μπορούν να καταφέρουν και αυτό διότι η ρήπανση διασχίζει μεγάλες αποστάσεις και περνά τα εθνικά σύνορα. Γι' αυτό και υπάρχει εδώ αυτός ο παράγωνο ενωσιακός και οπότε γι' αυτό και υποστηρίζουμε με τρεις τρόπους, με τρία μέσα ε, τη δράση των κρατομέλων. Πρώτα-πρώτα οι οδηγίες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Εκεί ορίζονται οι, οι, ελάχιστες υποχρεώσεις και έχουμε επίσης ε, το maximum της ε, συγκέντρωσης των βλαπτικών ουσιών στην ατμόσφαιρα και αυτό για πάρα πολλές ε, τοξικές ουσίες. Έχουμε επίσης την ε, οδηγία για τις οροφές, αν τα ανώτατα όρια δηλαδή των εκπομπών και έτσι θέλουμε να έχουμε κάποιους ε, καταλόγους για τις εκπομπές σε αιτήσια βάση όσον αφορά αυτούς τους μολυντές, τους παράγοντες μόλυνσης και τρίτον επίσης έχουμε και άλλα μέσα πολιτικής που θέλουμε να χτυπήσουμε τη μόλυνση στην πηγή και σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών. Σε αυτή την κατηγορία μέτρων έχουμε την νομοθεσία και την έγκριση τύπου για τα οχήματα και τις λεγόμενες, τους λεγόμενους ευρωκανόνες, Euro Norms, που και αυτό ε, νομίζω ότι είναι το βασικό θέμα που απασχολεί την Επιτροπή σας. Οπότε πάρα πολύ πρόσφατα είχαμε μια σφαιρική συνολική αξιολόγηση και ε, αυτό και θα συζητηθεί και είπαμε ότι αυτή η οδηγία για τα ανώτατα όρια εκπομπών ε, έχει απασχολήσει Κοινοβούλιο και Συμβούλιο και ήταν φιλόδοξος ο στόχος, δηλαδή το να μειωθεί η επίπτωση στην υγεία πάνω από 50% ε, μέχρι το 2030 σε σχέση 50% με το 2005. Είπε 48 το Συμβούλιο, 50 Επιτροπή και καλά κρατάνε διαπραγματεύσεις. Επίσης θα πρέπει να συγχαρώ την Τζούλι Γκέρλινγκ. Να τι έχουμε εδώ εκπροσωπήτη από την κόρη της εκεί στο έδρανο, η κυρία Γκέρλινγκ. Πρόκειται λοιπόν για κάποιον στρατηγικό στόχο, ο οποίος ε, αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Καθαρή Ατμόσφαιρα. Ο στόχος εκεί είναι το να υπάρχει συμμόρφωση μέχρι το 2020 το αργότερο. Και εάν έχουμε συμμόρφωση επομένω προς αυτές τις οδηγίες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, μέχρι το 2020, μέχρι το 2030 θα έχουμε μείωση στο 30% και η κατάσταση στην Ευρώπη δεν είναι ρόδινη. Οι οριακές τιμές του διοξιδίου του αζότου α, είναι πάνω από το, το, όριο ε, σε περισσότερο από 12 κρατημέλη, πάνω από 30 πόλεις. Και γι' αυτό και έχουμε αυτές τις υπερβάσεις που καταγράφονται από συσκευές της ε, κυκλοφορίας. Και επομένως ε, εκτίθενται οι Ευρωπαίοι ε, σε ρήπανση της ατμόσφαιρας. Και είπαμε ότι η πρόορη θάνατη που υπολογίζει η υπηρεσία περιβάλλοντος είναι πάνω από 70.000 ετησίως. Και αυτό παρά το ότι αυτά τα πρότυπα θεσπίστηκαν το 1999 και επέπρωτο να είναι δεσμευτικά από τον Ιανουάριο του 2012 και μετά. Όμως ήταν όλο ένα και πιο ξεκάθαρο ότι η συμμόρφωση όσον αφορά την συγκέντρωση του διοξιδίου του αζότου εξαρτάται από το τι εκπέμπουν ε, τα οχήματα που καίνε δίζελ. Και ακριβώς εδώ βλέπετε πού όλα αυτά κολλάνε ούτως ή στην στο έργο της Επιτροπής σας. Έχουμε τώρα ε, τα πρότυπα Euro 5, Euro 6 και είπαμε ότι υπήρξε παράταση τις θέσεις σε ισχύ κατά πέντε χρόνια και έφτασε ε, αυτή η πρόταση του 2014 για αυτές τις οριακές τιμές όσον αφορά το διοξείδιο του αζότου. Δυστυχώς όμως ε, τελικά ε, δεν έγινε αυτό και γι' αυτό τα οξύδια του αζότου από τα αυτοκίνητα που και είναι δίζελ έγινε ένας βασικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πώς θα τα θα περιορίσουν αυτές τις εκπομπές. Οπότε γι' αυτό και συνεργαζόμαστε ε, οι διάφορε υπηρεσίε και συνεργασίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά συνεργαζόμαστε και με άλλα θεσμικά όργανα και με τα κράτη-μέλη. Ο κ. πολύ σωστά μα είπε για το πρόγραμμα δράση, το σχέδιο δράση του 2020 και γιατί είπαμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε για τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη και τη βιομηχανία το πώς θα υπάρχει ασφάλεια, πώς θα είναι αυτή η βιομηχανία φιλοπεριβαλλοντική. Είναι κάτι το πάρα πολύ στρατηγικό βέβαια αυτή η βιομηχανία για την οικονομία μας. Απασχολεί 12 εκατομμύρια. Είναι επίση ο μεγαλύτερο κλάδο που δαπανά σε καινοτομία και έρευνα. Όμω υπάρχει και το θέμα τη κοινωνική ευθύνη από αυτή τη βιομηχανία, ούτω ώστε να, να μπορεί να ε, παράγει αυτοκίνητα περιβαλλοντικά. Ήδη από το 2012, μετά από εκτεταμένε διαβουλεύσει με τα κράτη-μέλη και με εννέα υπουργού εννέα επιτρόπους, εκπροσώπους ε, της ε, ΟΚΕ και όλους τους εμπλεκομένους αλλά ε, και συνδικά στελέχη αλλά και μη κυβερνικές οργανώσεις και χρήστες καταφέραμε σε κάποια συνενετικά συμπεράσματα. Οπότε το πρόγραμμα δράσης το οποίο τελικά εγκρίθηκε σε συμφωνία με όλους αυτούς κατέληξε στο ότι υπάρχει πρόβλημα με το διοξίδιο του αζότου και καταλήξανε στο ότι οι τωρινέ ε, διαδικασίες μέτρησης δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Και όλοι ξέραν επομένως ότι υπάρχει αυτό το χάσμα, αυτή η διαφορά μεταξύ των διαδικασιών μέτρησης και των πραγματικών εκπομπών. Οπότε και προτάθηκε ότι θα πρέπει να βρούμε ένα καινούριο κύκλο δοκιμών που να είναι πιο αντιπροσωπευτικός και να αντιστοιχεί στις ε, οριακές τιμές ε, του 2014 ε, του Euro 6 και να εφαρμόσουν αυτά από το, από το 2017. Συμφώνησε το Συμβούλιο, το Δευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συμφώνησε το 2013 κατόπιν της εξαιρετικής έκθεσης του κ. Προύστ και είπαμε μόνος ότι πρέπει να υπάρχει ένας κύκλος δοκιμών ε, πιο ακριβής. Οπότε διαμορφώθηκε συνένεση θεσμικών οργάνων και κρατών μελών και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Επίση, το 2010 συγκροτήσαμε την ομάδα έρευνα και ανάπτυξη, έκανα κάποια έκθεση και είχαμε επίση και την έκθεση JRC και έτσι μπορέσαμε να εισαγάγουμε στο σύστημα τι ε, μεταβολέ και να έχουμε έναν καλύτερο κύκλο δοκιμών, το RD και επίσης ε, όλα αυτά τα αγκάλιασε η βιομηχανία και υπήρξε ένσταση από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και θα έπρεπε εντατικά να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, να συμφωνήσουμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει συμμόρφωση και είπαμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει σε κάθε ε, περίπτωση να συμφωνήσουν με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικές επιτροπές για τα αυτοκίνητα και υπήρξαν επίσης και κάποια επιχειρήματα ε, από την βιομηχανία και λέγανε ότι θα, έπρεπε να υπάρξουν δοκιμές και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όλα αυτά καταγράφηκαν στην αξιολόγηση του 13. Οπότε θα έπρεπε στρατηγικά να κινηθούμε για να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση. Οπότε είχαμε διαδικασίε επί παραβάση, όπου δεν υπήρχε συμμόρφωση. Οπότε και έξι Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία ε, έλαβαν αυτή την επίσημη επιστολή όχληση για την παραβίαση, αλλά Αυστρία και Πολωνία επίση έλαβαν μια τέτοια όχληση και πρόκειται να ακολουθήσουν άλλες 7 χώρες που θα λάβουν τέτοια επιστολή, ότι δηλαδή ε, παρέβησαν τις οριακές τιμές του διοξιδίου του αζότου, αλλά επίσης δεν έκαναν και όσα προβλέπει η οδηγία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Όμως ήταν επίσης σημαντικό να υπάρχει κάποια συνέπεια και γι' αυτό τα κράτη-μέλη τα οποία ήταν λιγότερο πρόθυμα στην Τεχνική Επιτροπή να κινηθούν καλύτερα, οπότε και τους πιέσαμε για το RDE. Τώρα φτάσουμε στο Μάιο του 2015, οπότε έχουμε μια, θα έχουμε τέλο πάντων μια εφαρμοστική πράξη για να γίνουμε πιο φιλόδοξοι σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής, η οποία βέβαια κάπως απονευρώθηκε, αλλά, αλλά τώρα προχωρούμε και θα χρειαστεί να δίνουμε τις προσπάθειές μας. Τώρα είναι να σας αναφέρω τρεις δράσεις πολύ συγκεκριμένες, τις οποίες τώρα έχουμε αναλάβει. Πρώτα πρώτα θα συνεχίσουμε αυτές τις δικασίε σε παραβάση και εκτό από τα κράτη που σα ανέφερα που έχουν λάβει αυτή την επίσημη όχληση, πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλε τέτοιε ενέργειε, αν συνεχίσουν κάποια κρατημέλη, να περιβάλλουν τι ωρακέ τιμέ επίση. Δεύτερον, έχω γράψει σε κρατημέλη και του λέω ότι θα πρέπει να αναλάβουν δράση και έτσι να εξασφαλιστεί ότι οι υπερβάσει και η έκθεση του πληθυσμού θα πρέπει να συγκρατηθεί ε, μέχρι το 2020 κατά τρίτον ε, πώς θα να αξιολογήσουμε το, αν θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες. Παράδειγμα, να έχουμε κάποιους θελοντικούς μηχανισμούς, να έχουμε κάποια οχήματα χαμηλών εκπομπών ή πολύ χαμηλών εκπομπών. Τώρα, αυτό έγινε πριν, πριν έχουμε το σκάδο της Volkswagen και τέλος πάντων αυτός είναι ο βασικός μας ε, στόχος. Να επιταχύνουμε τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από αυτή την ε, πλευρά και από όλες τις πλευρές, ούτως ώστε να έχουν οι Ευρωπαίοι την ποιότητα ατμόσφαιρας που τους αξίζει. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρούνε Μέτσκερ. Γενικό Διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση για τι Κλιματικέ Αλλαγέ για να μα ενημερώσει μεταξύ άλλων και για τις δράσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις παρατυπίες ως προς τις ε, εκπομπές του άνθρακα. Ναι, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που προσκαλέσατε και τη Γενική μας Διεύθυνση, γιατί υπάρχουν και κλιματολογικές πτυχές σχετικές με τις εκπομπές του άνθρακα από ε, οχήματα με κινητήρα. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτήν την πρώτη συνεδρίαση να καλύψω τρία θέματα. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να περιγράψω ε, μια στιγμή επισκόπηση του ρόλου του συστήματος εγκρίσεως των ε, δοκιμών για διοξείδιο του άνθρακα και τη σχετική νομοθεσία οχημάτων που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα. Δεύτερον, θα ήθελα να αφαιρθώ στις αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών συνθήκων οδήγησης και των σχετικών εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα και της ε, τυπικής διαδικασίας και τρίτον, εν τέλει, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις δράσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις παρατυπίες ως προς τα δεδομένα στις, ε, τα σχετικά με τις εκπομπές οξύδου του άνθρακα που ανακοινώθηκαν το προηγούμενο φθινόπωρο από την ε, Volkswagen. Λοιπόν, αναφέρθηκε ο κανονισμός αυτός που αφορά τα οχήματα τα ισχύει από το 2009 και τα ελαφρά εμπορικά από το 2011. Οι δύο αυτοί κανονισμοί απαιτούν οι εκπομπές νέων οχημάτων που καταχωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ξεπερνούν συγκεκριμένους στόχους και ε, μειούνται ε, σύντο χρόνο. 130 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο για το 2015 και αντίστοιχα 95 γραμμάρια για το 2020 ήταν οι στόχοι που ορίζουν οι κανονισμοί. Εάν υπάρχει υπέρβαση ε, των στόχων αυτών, επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις συγκεκριμένα 95 ευρώ ανά γραμμάριο ε, διοξιδίου του άνθρακα κατά χιλιόμετρο για κάθε αυτοκίνητο που πωλείται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει αυτή την κύρωση. Τρεις περιπτώσεις έχουν ε, μέχρι στιγμή οδηγήσει σε κυρώσεις μέχρι ενό εκατομμυρίου, δεν σας αναφέρω τα ονόματα των συγκεκριμένων αυτοκινητοπαραγωγών. Ε, εν προκειμένου. Λοιπόν, ε, ορίζονται στόχοι, ορίζεται επαλήθευση συμμόρφωσης με τις δοκιμές, με τους τρέχοντες κύκλου δοκιμή, δοκιμών, NDEC, νέος κύκλος δοκιμών, που δεν είναι πια νέος, αλλά έχει μείνει το όνομα, New Driving Test Cycle, Σημαντικό επίσης είναι να αναφέρουμε τις ε, δράσεις για να αντιμετωπιστούν οι αποκλήσεις. Ο κύριος Πέτμακη αναφέρει ήδη ο ότι, αδίπο, ότι αυτές οι διαδικασίες των νέων δοκιμών του NDC e δεν είναι πλέον ε, ρεαλιστικές γιατί στηρίζονται σε τεχνολογία οχημάτων της δεκαετίας του 90. Όλο και μεγαλύτερη δηλαδή είναι η απόκληση μεταξύ αυτού που προτείνουν τα μέτρα με τις δοκιμές και τα αποτελέσματα των δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Λαμβάνονται υπόψη βεβαίως στην προετοιμασία της ε, νέας νομοθεσίας για στόχους διοξιδίου του άνθρακα αυτά τα δεδομένα και στις νέε νέες μας εκτιμήσεις. Δεν λαμβάνουμε αυτά τα στοιχεία σαν ε, ε, απόλυτα πίστα ως προς την πραγματικότητα, αλλά ε, κοιτάμε το σωρευτικό αποτέλεσμα για να διαμορφώσουμε τις προδιαγραφές. Στην, ε, και σε συμφωνία με τον UNICE και ανέφερε και ο κύριος Πετεμάκη τις ε, συνομιλίες. Έχουμε μια νέα διαδικασία προτείνει με το διοξίδιο του άνθρακα που θα αντικαθιστά την υφιστάμενη ενίδηση. Αυτή η νέα διαδικασία WLTP θα προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός, η δοκιμή δηλαδή για το διοξίδιο του άνθρακα και θα είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτική σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης με ευελιξία ως προς την διεξαγωγή των δοκιμών και ιδιαίτερα πιστεύουμε θα μειώσει αυτή η νέα μορφολογία των δοκιμών τις αποκλήσεις. Η Επιτροπή θα καταθέσει σύντομα και μας ενημερώσει ήδη ο κύριος Πέττεμακή τη σχετική πρόταση για την υλοποίηση ενός νέου καθεστώτος. Ε, πιστεύουμε ότι τα θεσμικά όργανα θα την ε, υποστηρίξουν την νέα αυτή πρόταση για να τεθεί το χειτροδυνατό σε ισχύ. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει μια νέα νομοθετική πρόταση για την περίοδο μετά τη 2020 με προδιαγραφές διοξιδίου του άνθρακα για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα που θα στηρίζεται σε νέα ε, και πιο αυστηρά πρότυπα WLTP με στόχο να αποφευχθούν πιθανές αυξήσεις των, και των αποστάσεων μεταξύ των αποτελεσμάτων των δοκιμών και των πραγματικών δεδομένων εκπομπών. Αυτό βέβαια με στόχο την εξυπηρέτηση της διαφάνειας και της ε, εμπιστοσύνης του καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή τα WLTP, αυτές, αυτή η δεύτερη φάση των ε, δοκιμών παραμένει σε εργαστηριακό επίπεδο και σε σχέση με άλλους ρυπογόνους, ε, είτε διοξίδιο του άνθρακα είτε μόνο οξείδιο του άνθρακα, δεν έχουμε προβλέψει για τις εκπομπές αυτές, δεν έχουμε εξασφαλίσει για τις εκπομπές αυτές ε, δοκιμή σε συνθήκες οδήγησης ε, επαρκώς και επιστημονικά γερή ώστε να ξέρουμε ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα. Ακολουθούμε φυσικά τις ε, συμβουλές των ειδικών, ε, επικοινωνούμε με επιστημονικά και πανεπιστημιακά ε, όργανα για να εξασφαλίσουμε στο δυνατόν καλύτερο υπολογισμό των εκπομπών στις συνθήκες οδήγησης. Τώρα, για τις ε, παρατυπίε τώρα συγκεκριμένα τη Volkswagen ω προ το διοξείδιο του άνθρακα. Ξέρουμε ότι στα τέλη του προηγούμενου έτου ανακοίνωσε η Volkswagen ότι μπορεί να υπάρξουν παρατυπίε και σε σχέση με τις εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα. Ανταποκρινόμενο σε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Volkswagen στην αλλά και από τι τοπικέ, από τι εθνικέ αρχέ πιστοποίησης να κοινοποιήσουν τον αριθμό και τα μοντέλα αυτοκινήτων που μπορεί να αφορά αυτή η ανακοίνωση, καθώς και το λόγο για τον οποίο υπάρχουν τέτοιου είδου παρατυπίες και άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχουμε λάβει απάντηση επί της ουσίας από την Volkswagen ή τις γερμανικές αρχές, άρα παραμένει εκρεμές το ζήτημα αυτής της απόκλησης. Κάθε χρόνο βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαληθεύει αν τηρούν τους στόχους διοξιδίου, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα η αυτοκινητοπαραγωγή και κάνουμε τις ε, σχετικές δημοσίευσεις για, το, για την επαλήθευση τήρηση των πρωτογραφών του 2014. Δεν κατέστη δυνατό να κάνει τη σχετική επαλήθευση σε σχέση με τον όμιλο Volkswagen η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι η σχετική της ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει στοιχεία για τη Volkswagen ακόμη ανακοίνωση το 2014, μόνο όταν μπορέσουμε να έχουμε καταληκτικά και πιστικά στοιχεία από τη Volkswagen και αντίστοιχα στι εθνικέ αρχέ, θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τι πληροφορίε και να καταλήξουμε σε μια απόφαση για το εάν ο όμιλο Volkswagen έχει τηρήσει τι δεσμεύσει σε σχέση και τη νομοθεσία σε σχέση με τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Καταλήγοντα, και δεν νομίζω να χρειάζεται να επαναλάβω αυτό που είπαν οι συνάδελφοι, είμαστε στη διάθεσή σα για να σα στηρίξουμε στην ε, περαιτέρω βελτίωση των προτάσεων. Ο στόχος μας, η στόχη μας είναι κοινή πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την επισκόπηση που μας προσφέρατε. Δύο γύρους ε, έρωτα αποκρίσεων προβλέπουμε. Με ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες και τους ηγητές βεβαίως σε πρώτη φάση, αλλά και μετά με μια διαδικασία catch the eye, όπου θα προσπαθήσω και εγώ να εξισορροπήσω την εκπροσώπηση των πολιτικών ομάδων. Ξεκινώ με τους δύο εισηγητέ όμως πρώτα. Κύριο Σπίτεχεμ, Σάλβα Μπίντεκεμ, Σάλβα Μπιντεγκάν και ο κύριος Γκερμπράντι μετά, αχ αυτά τα ισπανικά ονόματα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά το είπατε το όνομα μου, λέει ο κύριο Μπιντεγκάιν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τρεις ε, γενικούς διευθυντές για όσα μας εξήγησαν. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ήρθατε να μας τα εξηγήσετε και να απαντήσετε στις ε, ερωτήσεις που θα σας ε, θέσουμε. Ευχαριστούμε που είστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε την ουσία του προβλήματος όσο γίνεται με πιο διάφανο τρόπο. Κάποιες γενικές τώρα ερωτήσεις και πρώτους τρεις και σε μία συγκεκριμένη ερώτηση συγκεκριμένη τον κύριο Κάγεγα, όπως ε, είπατε κι εσείς, αρμοδιότητα βασική έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι, ε, από τη μία Επιτροπή και από την άλλη, άλλη αρμοδιότητα τα, τα κράτη-μέλη δεν υπάρχει ε, κοινή αρμοδιότητα. Γιατί είπατε για διαφορετικές αρμοδιότητες του καθενός. Δεύτερη ερώτηση. Μπορούν να κοιμούνται οι ήσυχοι οι Ευρωπαίοι, διότι τα μέτρα τα οποία εσείς εκπονείτε πρόκειται να παράσχουν κάποιες εγγυήσεις και ότι στο μέλλον οι αυτοβιομήχανοι ε, να συμμορφωθούν κάτι άλλο για το παρελθόν κάνατε στο παρελθόν αρκετά για να αποφύγουμε ε, την χρήση των επίμαχων και των επιλήψιμων συσκευών. Επίσης, οι επιπτώσεις των μέτρων σας, ποιες θα είναι όσον αφορά την απασχόληση, γιατί ο, αυτός ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος. Άρα με αυτά τα μέτρα τα οποία εκπονείται, μήπως είναι δυνατόν να δώσουν μια όθηση στην απασχόληση στον οικονομικό αυτόν κλάδο. Συγκεκριμένως για τον κύριο Καγιάχ μας αναφέρετε εσείς αυτό το σχέδιο δράσης, το CARS 2020. Και αν δεν κάνω λάθος είπατε ότι εντατικά ε, το επεξεργάζεστε. Ξέρετε ότι με αυτό το πρόγραμμα, αυτό το πλάνο ε, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη διαφορά μεταξύ των μετρουμένων ε, εκπομπών και των πραγματικών. Επίσης, ξέρετε ότι εμείς επιψηφίσαμε εκείνη την έκθεση και όλοι που επιψηφίσαμε είπαμε επιλέξει ότι ναι θέλουμε να υπάρχει αυτός καινούργιος κύκλος δοκιμών και να υπάρχουν τέτοιου είδους ε, δοκιμές που να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης και ότι όλα αυτά αμελητή θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή. Οπότε, φαντάζομαι πάνω να πει ότι γνωρίζαμε όλοι το πρόβλημα. Και αφού το γνωρίζαμε εμείς, φαντάζεστε ότι θα υπήρχε κάποιος από εμά που να κάτσει και να ζητήσει τη συγκρότηση αυτής της ε, Εξεταστικής Επιτροπής. Κύριε Χέρμπραντ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, τηρήστε το όριο των δύο λεπτών. Ευχαριστώ πολύ. Και ιδιαίτερα σε ευχαριστώ τις τρεις γενικές διευθύνσεις που έχουν εδώ εκπροσώπηση και έτσι δίνουν και το αναρκτήριο λάπτισμα για τη δουλειά αυτής της Επιτροπής. Έχω τις έξι ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την ίδια την Επιτροπή εν γέννη Ακούσα σαφείς και περίφραστες δηλώσεις ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να επαναληφθεί κάτι τέτοιο και όλα αυτά. Συμφωνώ απολύτω. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο το Κοινοβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Και φαντάζομαι ότι και η Επιτροπή η ίδια διερευνά από πλευρά τη γιατί συνέβη ό,τι συνέβη. Συνεργάστηκαν σωστά οι γενικέ διευθύνσει μεταξύ του ήταν επαρκής η πίεση που άσκησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν υπάρχει μια εξεταστική διαδικασία η Επιτροπή μες στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να το ξέρω. Εάν δεν υπάρχει θα ήθελα να ξέρω και γιατί δεν υπάρχει. Και ίσως εάν υπάρχει αυτή η Επιτροπή μπορούσατε να μας δώσετε τα στοιχεία στα οποία έχει καταλήξει και τα πορίσματά της. Επίσης για, την, ε, για τις αρχές εποπτείας αγοράς ο κύριος Πατμακή έκανε μια διάκριση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, ότι δηλαδή η Ευρώπη έχει ένα πολύ πιο ε, πρόημο σύστημα υποπτήρες αγοράς, ενώ οι ΗΠΑ Πολιτείες ε, παρεμβαίνουν εκ των υστέρων. Ε, εγώ πάντως βλέπω ότι οι αρχές υποπτήρες αγοράς μπορούν να ελέγξουν αυτοκίνητα. Είναι το λεγόμενο in-service conformity tests, τα οποία ήδη έχουν ε, ε, μπει στην αγορά. Μπορείτε λοιπόν να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω πού έγκυνται αυτές οι διαφορές. Έχουν αυτές οι δοκιμές ε, πραγματοποιηθεί. Εάν δεν πραγματοποιήθηκαν, γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν. Και μήπως μπορείτε να μας πείτε και δύο λόγια για αυτές τις ε, ενδοϊπηρεσιακές επαληθεύσεις συμμόρφωση όπως ονομάζονται in service conformity tests παρακαλώ ο κύριος Κίσεκε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πράγματι πολύ θετικό το ότι έχουμε εκπροσώπους και από το περιβάλλον και από την ανάπτυξη και από τις κλιματικές αλλαγές ε, εδώ. Βεβαίως αυτή η δουλειά ξεκινάει σήμερα, πρώτη μέρα, πρόκειται για μια δωδεκάμινη εντατική εργασία που ξεκινάει σήμερα. Πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει πολύ επικοδομητικά και εμείς ως πολιτικοί θα πρέπει να διαρωτηθούμε εάν, μια και το ανέφερε και ο κύριος Μέτσκερ, έχουμε ενδεχομένως ε, αφήσει σε μεγάλο, βαθμό στα χέρια της αυτοκινητοβιομηχανίας το στόχο της μείωσης των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Και επίσης υπάρχει και το ζήτημα των οξυδίων του αζότου ε, μήπως θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια επιτάχυνση των διαδικασιών. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να υπερηφανευόμαστε γιατί έχουμε ε, βοηθήσει στην ταχύτερη πρόοδο των εργασιών και για τα έλαφρα εμπορικά οχήματα 3,5 χρόνια. Ε, πώς μπορούν λοιπόν να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες ε, και με τη βοήθεια φαντάζομαι των εμπειρογνωμόνων γιατί ο στόχος μας είναι όντως κοινό. Πέραν των εργαστηριακών τιμών δηλαδή πρέπει να μπορούμε να κάνουμε ε, μέτρηση και των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Επίσης, η διαπίστωση των παραβάσεων έλαβε χώρα σε στι ΗΠΑ, πράγμα το οποίο βρίσκω πολύ λυπηρό, δεν έλαβε χώρα στην Ευρώπη. Τι έχει κάνει λοιπόν συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε απόκληση μεταξύ των ε, εργαστηριακών και πραγματικών ε, δοκιμών και γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ω προ τα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ΗΠΑ. Εντάξει, υπάρχει το ζήτημα τη έγκριση πριν από τη θέση σε ε, κυκλοφορία των οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε περισσότερο δρούν μετά τη θέση κυκλοφορία, αλλά θα έπρεπε να βελτιώσουμε τι σχετικέ διατάξει, γιατί ε, πρέπει να υπάρχει ουσιαστική βελτίωση. Και ξέρετε ότι θα έχουμε να κάνουμε μία έκθεση για το τέλο του χρόνου και περιμένουμε συγκεκριμένε προτάσει ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κύριο Ντόνς Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Και σε ευχαριστώ όλου που είστε εδώ. Είναι καλό το ότι έχουμε ένα ευρύ φάσμα από τη δουλειά της Επιτροπής. Βεβαίως, στη διάρκεια αυτής της εξεταστικής Επιτροπής θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα πραγματικά περιστατικά. Τι συνέβη και πότε. Με χαρά βλέπω ότι δόθηκαν εξηγήσει προς την γραμμή του χρόνου αυτής της ε, διαδικασίας αλλά κάποια πράγματα με μπέρδεψαν λίγο από τις δηλώσεις που άκουσα και θέλω διευκρινήσει. Η νομοθεσία λοιπόν 2007 με την υλοποίηση της να ξεκινά το 2009 αλλά κάποιοι που υπόθηκε quite soon after, σύντομα μετά είπατε εσείς. Και αυτό τα είχα εξηγεί και ε, μάλλον ε, δείχνει ότι η Επιτροπή σύντομα μετά αντελήφθη ότι υπήρχαν αποκλήσεις μεταξύ εργαστηριακών δοκιμών και ε, αποτελεσμάτων δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες. Αλλά δεν προχωρήσατε σε ε, αντιμετώπιση του προβλήματος και μετά το 2012 μόνο θεσπίστηκε η σχετική επιτροπή. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η καθυστέρηση μετά την ε, συνειδητοποίηση των προβλημάτων των σχετικών με, την, με τα πραγματικά δεδομένα και την ανάληψη μέτρων της επιτροπής που και πάλι δεν έχουν τελείως ξεκαθαρίσει. Και επίσης θα ήθελα πιο πολλά στοιχεία σε σχέση με την, τη CMB, Τεχνική Επιτροπή δηλαδή. Ποιος συμμετέχει στην Επιτροπή αυτή. Θέλουμε λεπτομέρειες για τα μέλη της, τις συνεδριάσεις της, τις αποφάσεις που ενδεχομένως επηρεάζει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. την ε, ενδεχόμενη ενημέρωση ή ε, νέα στοιχεία που μπορεί να προκύπτουν όχι μόνο από αυτά που σα λένε τα κρατη αλλά από τη δουλειά ιδιαίτερα αυτή τη Επιτροπή. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο και κύριο που τηρείτε και το χρόνο σα, ο κύριο Χένκελ, CR. Τρεις ερωτήσεις μόνο. Πρώτον, και παρουσία της Επιτροπής. Ε, έχετε και εσείς την εντύπωση, όπως εγώ, ότι συγχέονται δύο διαφορετικά θέματα, θεματολογίες προβλημάτων. Καταρχάς, ε, τα αποτελέσματα ε, των εργαστηριακών δοκιμών σε σχέση με τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης αφενός, αλλά αφετέρου ένα άλλο πρόβλημα που είναι η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Volkswagen συγγνώμη, να στρεβλώσει τα αποτελέσματα με το λεγόμενο defeat device. το μηχανισμό παράκαμψης γιατί εμφανίζονται αυτές οι διαφορές, γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και φαίνεται από το μαθαίνω ότι και η γερμανική κυβέρνηση διαπιστώνει πως το πρόβλημα περιορίζεται μόνο στη Volkswagen και ότι δηλώνει πως δεν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα με άλλους ε, κατασκευάστες αυτοκινήτων. Υπάρχουν ε, σχετικά πορίσματα, δικές σας, ε, δικά σας ευρήματα. Ευχαριστώ. Κύριος Ροσφόρ Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους τρεις αναπληρωτές γενικούς διευθυντές. Ξεκινώ λέγοντα τρία πράγματα Σα σας άκουσα. Πρώτον, λέμε όλοι το ίδιο πράγμα, δηλαδή πώ είναι δυνατόν να το αντιλαμβάνονται στι ΗΠΑ και να μην το έχουν αντιληφθεί στην Ευρώπη ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό μα προβληματίζει όλου, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Και η δική μου η οπτική, και με αυτόν τον τρόπο σα ρωτάω καιρό. όλοι γνωρίζαμε εδώ και χρόνια ότι δεν ήταν οι πραγματικές επιδόσεις των αυτοκινήτων ε, αυτές οι οποίες αναγράφονταν. Μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν έχουν μόνο στις ΗΠΑ. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσάς δηλαδή, τόσα χρόνια οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν σας έλεγαν ότι δεν, δεν είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα αυτές οι τιμές. Τι τις κάνατε αυτές τι παρατηρήσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τις αγνοήσατε, τις παραπέμψατε στις καλένδες, τι κάνατε. Δεύτερον, Λέγεται ότι υπάρχει αποκέντρωση, αρχή της επικουρικότητας, στα 28 κράτη-μέλη στην Ευρώπη κτλ. κτλ. Εξηγείται το φαινόμενο. Μα αυτό μας κάβει ακόμα περισσότερο το λάκκο. Γιατί είναι σαν να μας λέει το ευρωπαϊκό σύστημα, σύν τα 28 ε, εθνικά συστήματα, 29 το, το όλων, ήταν σε απόλυτη ανικανότητα να ε, διαπιστώσουν ένα πρόβλημα το οποίο μας αφορά το μεγαλύτερο κατασκευαστή αυτοκινήτων της Ευρώπη Και τρίτον, δεν αναφέρθηκε εξ αρχή. Ο καταναλωτή όμω, ο Ευρωπαίο καταναλωτή ήταν το κύριο θύμα αυτή τη ε, υπόθεση αυτού του σκανδάλου. Και για λόγου περιβαλλοντικού, αλλά και ω καταναλωτή. Γιατί αγόρασε προϊόν το οποίο τον εξαπατά. Έχει απατηλέ δηλώσει. Έτσι λοιπόν, εσεί τι λέτε σήμερα ω Επιτροπή στον καταναλωτή, πώ θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά, στην ενιαία αγορά του καταναλωτή και για προϊόντα σημαντικά όπως τα οχήματα με κινητήρα. Δεν είναι δουλειά μιας επιχείρησης μόνο ή του ε, κατασκευαστή αυτοκινήτων αν προκειμένου να αναλάβει αυτό το καθήκον. Γιατί στη τελευταία ανάλυση εσείς η Επιτροπή, εμείς αλλά πάνω απ' όλα εσείς είστε ο θεματοφύλακας και των θεμητών και νομίμων δικαιωμάτων του καταλωτή, ο οποίος θεωρεί ότι εσείς τον προστατεύετε και επαχρυπνείτε. Ευχαριστώ κύριε Κίλλονεν. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους τρεις καλεσμένους μας. Το Joint Research Center Δηλαδή, η Εσωτερική Υπηρεσία Ερευνών τη ευρωπαϊκή επιτροπή είχε πει το 2013 ότι οι συσκευέ παράκαμψη που χρησιμοποιεί Volkswagen αλλά και άλλε εταιρείε μπορούν να παραποιήσουν τα αποτελέσματα μετρήσεων εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, δεν θα έπρεπε να είχε λάβει πιο σοβαρά υπόψη στη γνωμοδότηση αυτή της JRC και δεν θα έπρεπε να είχε αναλάβει πιο προσήκουσα δράση γιατί νομίζω ότι από το 2013 μέχρι τη στιγμή εκείνη που λάβαμε τις πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν πολλά χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αντιλαμβάνουμε δράση πολύ πιο γρήγορα. Αυτό θα πρέπει να είχαμε κάνει στο παρελθόν. Πρώτο ερώτημα αυτό. Δεύτερον, αν αναλύσουμε το εφιστάμενο σύστημα επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, υπάρχει κάποια ένδειξη ότι το σύστημα RDC ουσιαστικά συνδέει τους ίδιους κατασκευαστές με αυτό το σύστημα μέτρησης των εκπομπών, έτσι να μπορούν τελικά να το επηρεάζουν. Η κυρία Ντάλη και το λόγο ξενόματος των Πρασίνων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω η παρουσία εδώ σήμερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποτελεί ένα μιας πολύ επικοδομητικής και ειλικρινής συνεργασίας για το ζήτημα αυτό, γιατί πρέπει να χυθεί άπλετο φως σε όλους αυτούς τους παράγοντες που δίγησαν σε αυτό το σκάνδαλο. Αν πραγματικά θέλουμε η διαφάνεια να αποτελέσει πάγιο κανόνα, θα πρέπει να εξαφανίσουμε οποιαδήποτε κενά νομοθετικά τα οποία επιτρέπουν τελικά τη μη διαφάνεια. Το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό. Κύριε Πελτομάκη από τη Γενική Διεύθυνση Growth, σας ευχαριστώ καταρχάς που είστε εδώ πέρα. Πριν από ένα χρόνο, ο κύριος Στένερζε από την υπηρεσία σας, μία Κυριακή, πήγε και συνάντησε τους LCOA, το λόμπι δηλαδή της αυτοκινητοβιομηχανίας, και μαζί συζήτησαν τις ρηπογόνες αυτές εκπομπές. Όπως λέγεται στο Corporate Europe Observatory, νομίζω ότι θα πρέπει να καταγράφονται όλες οι επαφές που έχουν όλοι οι εξωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με οποιαδήποτε λόμπι. Σας ζητά λοιπόν το παρατηρητήριο αυτό το οποίο ανέφερα να επιβεβαιώσετε ότι όντως έγινε η επαφή αυτή του φυσταμένου σας με εκπροσώπου ε, του λόμπι τη αυτοκινητοβιομηχανία. Δύο απόπειρε γίνανε, δεν δώσετε καμία απάντηση για ποιο λόγο τέτοια σιωπή, για ποιο λόγο τέτοια συγκάλυψη απέναντι σε επαφέ αυτέ που ενδεχομένω να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και με συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Ελπίζω ο κύριο Στένερζε να έρθει εδώ πέρα στην εξαιρετική μα επιτροπή προκειμένου να μα πει όλη την αλήθεια για το ζήτημα αυτό. Δεύτερον, αν δούμε τον, ε, το δημόσιο μητρό βλέπουμε ότι υπήρχαν 13 συναντήσεις, 13 το αριθμό συναντήσεις μόνο και μόνο το 2015 με την ΣΕΑ. Ε, υπάρχουν πρακτικά από τις συναντήσεις αυτές, είναι δημόσια τα πρακτικά αυτά, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα πρακτικά, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα ζητήματα τα οποία συζητάτε κάθε φορά και ποιες θα οι επόμενες, οι μελλοντικές προβλεπόμενες συναντήσεις με αυτό το λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας. Κύριε Καλέχα, τώρα απευθύνομαι σε εσά. Είστε ο εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο. Στο παρελθόν συμμετείχατε και εσεί στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη, η οποία δεν ονομαζόταν τότε DG Growth αλλά DG Enterprise για τι επιχειρήσει. Πώ αλλάζουμε τόσο εύκολα βασικά ιδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να εκπροσωπούμε δηλαδή τη μια μέρα την αυτοκινητοβιομηχανία και την επόμενη μέρα την υγεία των καταναλωτών. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το είπατε κι εσείς ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλήσεις ανάμεσα στις εργαστηριακές δοκιμές και τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Για ποιο λόγο δεν έγινε τίποτα άλλα αυτά τα χρόνια, ενώ είχατε εντοπίσει ότι υπήρχε, υπήρξε τέτοια μεγάλη απόκληση. Και ο αρμόδιος επίτροπος τότε για το περιβάλλον είχε έρθει σε επαφή με τον κύριο Ταγιάννη, ο Τέτνικ, είχε έρθει σε επαφή με τον κύριο Ταγιάννη. Συγγνώμη, πρέπει να τα πω όλα αυτά, γιατί πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Για ποιο λόγο συγκαλύφθηκε και αυτό και δεν υπήρχε καμία ενημέρωση όσον αφορά τις επαφές αυτές. Κυρία Ντάλη, πρέπει όλοι, όλοι να τηρούμε το χρόνο αγόρευσης. Είναι η πρώτη μας συνάντηση, θα ακολουθήσουν και πολλές άλλες. Εξ ονόματος του EFDD, κυρία Εύη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις θα υποβάλω, πολύ συγκεκριμένες. Πρώτα πρώτα τι γίνεται με τα κίνητρα. Τα κίνητρα, τις επιδοτήσεις, ενισχύσεις. Με ποιο τρόπο εσείς εξασφαλίσατε ότι θα υπάρξουν κίνητρα ούτως ώστε στην αγορά να πιάσει τόπο ε, το, το, το μέτρο αυτό για τα πρότυπα ευρώ και οπότε τελικά να γίνουν σεβαστές οι, παρά, οι παράμετροι όπως έχουν τεθεί για τις εκπομπές. Επίσης, η DG Crow σε πρώτη φάση θεωρείτε ότι αυτές οι εκπομπές έχουν ξεπεράσει εκείνες που παρατηρούνται και καταγράφονται σε πραγματικές συνθήκες στον δρόμο. Δεν νομίζετε ότι έχει, έχει λάβει σοβαρό χτύπημα η ιδέα το μέτρο του Euro 6. Οπότε πώς θα μπορούσαμε να πετύχουμε τους στόχους που μέχρι τώρα κανένα δεν έχουμε πετύχει. Επίσης για τις παραβάσεις. Έχουμε όλα αυτά τα κρατημέλη τα οποία ακριβώς έχουν πέσει σε παράβαση και έχουν φτάσει σε διπλάσιες ε, τιμές σε σχέση με αυτά που προβλέπονται στις πραγματικές τιμές του δρόμου. γιατί μια σύγχυση, οπότε τι θα γίνει με αυτές τις παραβάσεις. Πώς θα μπορούσε να, ε, να αντιδράσει ε, Κρατό μέλος σε αυτή τη ε, διαδικασία παραβάση. Ευχαριστώ πολύ, πρώτος. Μίλησαν από σε όλες τι πολιτικές ομάδες. Ε, οι εκπρόσωποι τώρα έχουμε τους ε, τρεις τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κανονίστε τώρα πώ θα απαντήσετε. Είναι πολύ δύσκολο να μοιράσουμε τι ερωτήσεις. Μερικές απευθυνόταν συγκεκριμένα σε κάποιον από εσά, μερικές επικαλύπτονται και έχουμε και κάποιες ερωτήσεις προς το της Επιτροπής σε σχέση με αυτά που είχατε προηγουμένως κάνει. Αν μπορείτε περιοριστείτε κύριε Πελτομάκη πρώτος εσείς να απαντήσετε τηλεγραφικά σε ένα πεντάλεπτο. Ε, Πρόταση. Ερωτήσει από τον κύριο Μπιντεγκάιν. Ο διαχωρισμός της αρμοδιότητας. Προ, προ, να σας πω ότι εμείς νομοθετούμε και τα κράτη-μέλη υλοποιούν και εφαρμόζουν. Και εμείς μετά παρεμβαίνουμε με τη διαδικασία επί παραβάση. Κάτι το οποίο βγήκε και από άλλες ερωτήσεις. Χρειάζεται για να προβούμε σε αυτή τη διαδικασία η παραβάση να έχουμε ξεκάθαρες ενδείξεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις ότι υπήρξε υπέρβαση των οριακών τιμών, όπως ορίζει ο νόμος. Και φυσικά επικαλούμαστε και τα τεστ που προβλέπει η νομοθεσία. Έτσι μπορούμε να μετρήσουμε το αν υπάρχει συμμόρφωση ή όχι. Και βεβαίω θέλουμε να αναβαθμίσουμε αυτές τις διαδικασίες, να τις βελτιώσουμε. Και έτσι να αποπτεύσουμε την αγορά. Βεβαίω υπάρχουν αδύνατα σημεία και μειονεκτήματα σε αυτή τη διαδικασία εποπτεία τη αγορά. Γενικότερα για την αυτοκινητοβιομηχανία και όχι μόνο για τις εκπομπές. Αναφέρεται και τις ε, νομένες Πολιτείες και είπαμε ότι περισσότερο προσέχεται η εποπτεία της αγοράς στη ΣΥΠΑ παρότι εδώ. Εδώ έχουμε κυρίως την, ε, την έγκριση τύπου και αυτό εξηγεί γιατί στη ΣΥΠΑ ανακαλύψαν τι γίνεται. Και βέβαια υπήρχαν βέβαια κάποια ευρήματα από την ε, υπηρεσία περιβάλλοντος την Ευρωπαϊκή και κατόπιν αποδέχθηκε τις κατηγορίες η Volkswagen. Τώρα όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης και τους καταναλωτές. Εμείς επεξεργαζόμαστε λύσεις για αυτά τα σημεία και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο αυστηροί, να λάβουμε υπόψη δηλαδή τους ε, στόχους όπως περιβάλλον και ασφάλεια. Και όλα αυτά όμως εξασφαλίζοντας ότι θα είναι πρωτοπόρες οι βιομηχανίες μας στην παγκόσμια κούρσα. Πρωτοπόρες και όχι ουραγή. Και έτσι προβλέπονται σχετικές απαιτήσει για τα οχήματα. Βέβαια έχουμε και κάποιες πολιτείες στη ΣΥΠΑ που έχουν ακόμα πιο αυστηρές προδιαγραφές Θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική η βιομηχανία μας και τέτοιου είδου λύσεις θέλουμε να εξευρεθούν σε σχέση με τι χρειάζεται παγκοσμίω, γιατί το θέμα της μείωσης των εκπομπών είναι θέμα επικαιρότητα και σε ΙΠΑ και σε Κίνα. Γι' αυτό σας λέω. Ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα καινοτομήσουμε, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε πολύ αυστηροί στα προπετούμενα που θέτουμε, αλλά τελικά να βρούμε και κάποια λύση η οποία θα βοηθήσει την απασχόληση αλλά και την ανταγωνιστικότητα. Άλλη ερώτηση. Αυτό το δημοσίευμα σε εφημερίδα που είπατε κάποια κυριακάτικη δημοσίευση του Ιανουαρίου αυτή η συνάντηση που είπατε δεν έγινε τότε είχε προηγηθεί ή ακολούθησε τέλος πάντων εμείς πάντα με τους εμπλεκόμενους και με την ΑΣΕΑ όπου αναφέρει το δημοψήφισμα συλλομιλούμε ανοιχτά με διαφάνεια Αυτοί δημοσίευσαν και κάτι φωτογραφίες από την ΑΣΕΑ και υπονοούσαν ότι υπάρχουν κάποια deal μεταξύ των εμφανιζομένων ε, στο δημοσίευμα. Όχι, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Βεβαίως και συζητάμε. Και θέλουμε να έχουμε τη γνώμη όλων. Αλλά όλοι μας οι συνεννοήσεις γίνονται με ξεκάθαρους κανόνες και όσο αυτές τις σχέσεις με τα λόμπι. Όσο γίνεται περισσότερο είμαστε ανοιχτοί σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθούμε. Άλλε ερωτήσεις για να δω. Ο Επιτροπή δεν έχει συγκροτήσει κάποιο είδου ε, εξεταστική επιτροπή δεν έχει κάνει κάποιο έρευνα. Προετοιμαζόμαστε να βοηθήσουμε τη δική σας εξεταστική επιτροπή. Να συντονιστούμε, να συμφωνήσουμε για τις ακολουθητές διαδικασίες και χάρη σε εσά τώρα γίνονται μέχρι των υπηρεσιών μας διαβουλεύσεις επί τη βάση των όσων εσείς προτείνετε και συζητάτε να καταλάβουμε όλοι τι έγινε, γιατί έγινε και από ποιον. Και θα σας δώσουμε ό,τι πληροφορίες θέλετε. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, σας ε, βεβαιώνω ότι η σύγκριση τα ξέρων και των διατάξεων που ισχύουν στις ΗΠΑ και την Ευρώπη θα είναι αντικείμενο μιας από τις ακροάσεις που θα γίνουν πριν από τις θερινές διακοπές. Το ξεκίνημα μόνο είναι και θα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Παρακαλώ εσείς. Πρόεδρε, ευχαριστώ και θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις στα όσα δεν κάλυψε ο κύριος Πέκτομακή. Ξεκίνησα από τον κύριο Σάλβα για το ΚΑΡΣ 2020. Αυτή η ομάδα εργασία. Εκεί συμμετέσχουν κρατημέλη, βιομηχανία, με κυβερνικέ οργανώσεις και κατέληξαν στο εξή ότι τα τεστ δεν αντιπροσωπούσαν πραγματικές τιμές. Αναζητήθηκε λύση και ζήτησαν να υπάρξει έντονη συνεργασία και εντατική της Κομισιόν και των κρατών μέλων. Δεν φτιάξαμε ερευνητική επιτροπή, όμως προτεραιότητα ήταν να φτιάξουμε ένα καινούργιο σύστημα στην Ευρώπη λειτουργικό, που έτσι να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες των σημερινών τεστ. Αυτό το ξέραν όλοι. Ότι δεν είχαμε πραγματικές ρεαλιστικές τιμέ. Άρα θέλαμε σύστημα λειτουργικό, αποδοτικό, να αλλάξει το σύστημα να μπορέσουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε απάτη. Ακριβώς όπως είπατε πολύ εξημών. Έπρεπε αυτό να καταφέρουμε. Δεν έγινε. Να, η έρευνα που οφείλει να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις. Οπότε έτσι θα γίνει. Το καινούργιο σύστημα θα καλύπτει αυτά τα συστήματα φορητά συστήματα εκπομπών, ούτως ώστε να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις. Δεν είχαμε τέτοιο σύστημα στα αυτοκίνητα. Α, γι' αυτό φτάσαμε εκεί. Από το 2017 θα υπάρχουν αυτές οι συσκευές στα αυτοκίνητα και αυτό είναι η καλύτερη εγγύηση ότι δεν θα ξαναγίνουν τέτοια πράγματα. Βεβαίως, αυτά συνέβησαν και αποτελούν γεγονός που δεν θα θέλαμε να είχε συμβεί. Όμως υπήρχε και ένα δεύτερο αδύνατο σημείο και δυσκολία. Το ότι εμείς προβλέπουμε κάποιους κανόνες, θεσπίζουμε, αλλά τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν και έχουν ε, την πιστοποίηση και την έγκριση τύπου. Δεν έχουμε αρκετούς υπαλλήλου για να τα ελέγξουν όλα αυτά. αυτή την πιστοποίηση, την έγκριση, την ομολογκασιόν τα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν τι γίνεται και πώς εφαρμόζεται το σύστημα της εγκρίσης τύπου. Ε, μια άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Γιατί είναι τόσο περίπλοκα τα συστήματα, τα σχετικά στην Ευρώπη και η νομοθεσία, η σχετική. Μα δεν πρόκειται για μία χώρα, είμαστε 28 χώρες. Το προβλεπόμενο σύστημα βασίζεται σε πρωτοβουλία της ε, Κομισιόν Έχουμε τη σχετική επιτροπή. Θα πρέπει στην επιτροπή να πριτανεύσει η ειδική πλειοψηφία που είναι δύσκολο. Θα πρέπει όλες οι συναρμόδιες επιτροπές να εξεύρουν ειδική πλειοψηφία. Αλλιώς κάποιο μέτρο δεν μπορεί να περάσει. Θα πρέπει να περιμένουμε τρεις μήνες επίσης να περάσει η πρόταση από Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Ε, έτσι κινούμεθα και εμείς πρέπει να τηρήσουμε το τι προβλέπεται. Αλλά τώρα αλλάζουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Άλλη ερώτηση. Ποιοι συμμετέχουν στην Επιτροπή για τα αυτοκίνητα. Πρόσωπο, τα κράτη-μέλη είναι κανονιστική, ρυθμιστική αυτή η Επιτροπή και διέπεται από την Επιτροπολογία. Χένκελ. Απαντήθηκε τα σχετικά με τις διαφορές ε, όσον αφορά και είπε και η πρόταση θα γίνει ad hoc ε, Επίσης ο κύριος Ροσφόρ έλεγε τι απάντησε μη κυβερνικές οργανώσεις η Επιτροπή. Τους είπαμε ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές και εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε το σύστημα ότι υπάρχει αυτή η απόκληση μεταξύ πραγματικότητας και, και, και μετρήσεων. Η απόκληση δεν πάει να πει ότι υπάρχει εξαπάτηση. Άρα με το νέο σύστημα αυτό ελπίζουμε ότι θα έρθουν αυτές οι διαφορές με αυτό το σύστημα portable emissions. Κύριε Κιλώνα, ρώτησε γιατί δεν παίρνει πιο σοβαρά τα συμπεράσματα της JRC. Φυσικά και πήραμε στα σοβαρά τα όσα διατύπωσαν στην έκθεση. Αυτό αφορούσε η έκθεση, το πώς θα εξυπηρεστεί το πρόβλημα, πώς θα έχουμε καινούριο σύστημα. Να βάλουμε αυτό το Portable Emission System, το PEM, στα αυτοκίνητα. Αυτή ήταν η πρόταση. Κύριε, θα, θα είμαι επίση ειλικρινή μαζί σα, Από το 1986 εργάζομαι και ω ε, υπάλληλο και έχω περάσει από πολλές θέσεις και ξεκίνησα από την νομική υπηρεσία και το πρώτο που έκανα ήταν να σύρω τη χώρα με ενώπιον του δικαστηρίου. Σε μεταφορέ, σε ενέργεια έχω εργαστεί. Στη διεύθυνση βιομηχανία, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τώρα είμαι στη διεύθυνση για το περιβάλλον. Νομίζω ότι η κινητικότητα είναι κάτι το θετικό να ενθαρρυνθεί και άλλοι όπως εγώ έχουν ακολουθήσει τέτοια διαδρόμια. Και εγώ όπου και εργαζόμαστε υπεραμεινόμεθα του, των συμφερόντων της Ευρώπης. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Μέτσκερ, τώρα εσείς έχετε το λόγο. Ναι, και θα είμαι σύντομος, κυρία Πρόεδρε γιατί οι συνάδελφοί μου έχουν, ε, με έχουν καλύψει, απάντησαν στι περισσότερες ερωτήσεις. Υπήρχε μία ερώτηση βέβαια που είχε να κάνει με εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα και με τα αντιζαλοκίνητα αυτοκίνητα. Και νομίζω ότι αυτό συνδέεται και μετά όσο είπε ο κύριο Χένκελ. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα δύο αυτά ζητήματα. Από τη μία πλευρά έχουμε διαφορέ ανάμεσα στις εργαστηριακές δοκιμές και τις δοκιμές μέτρησης σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και νομίζαμε ότι μπορούσαμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά, αλλά δεν είχαμε καταλάβει ότι στην περίπτωση Volkswagen υπήρχε και ένας ακόμα παράγοντας, οι συσκευές παράκαμψης. Τώρα, υπάρχουν και άλλες όμως εταιρείε οι οποίες καταφέρνουν και πετυχαίνουν με διάφορες τεχνικές λύσεις συγκεκριμένα επίπεδα εκπομπών, όπως για παράδειγμα για τις ρηπογόνες ουσίες στην ατμόσφαιρα, για τις οποίες υπάρχουν πάλι τεχνικές συσκευές που βοηθούν κάποιες εταιρείες να πετυχαίνουν τα απαραίτητα μέτρα. Βέβαια, αν μια εταιρεία τώρα θέλει να χρησιμοποιήσει συσκευή παράκαμψης, μπορεί να το κάνει, προκειμένου να δείξει ότι τα οχήματά της συνάδουν συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρος. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ο Ιβάν Πέλετ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. πόσο, ένα λεπτό, μισό λεπτό, ενάμιση. Δεν θυμάμαι τι είχατε πει στην αρχή. Ε, αν μπορείτε να είστε όλοι κάτω από τα δύο λεπτά θα τα καταφέρουμε έτσι. Πρόεδρε, ευχαριστώ τεχνική ερώτησή μου ε, και προς τον κύριο Ρέτσικερ και τον κύριο Καλέχα και ευχαριστώ σας βεβαίως που ήρθατε για την αξιολόγηση συνεπειών ε, για το Euro 5, Euro 6 το 2007. Τα διαβάσαμε, τα ξαναδιαβάσαμε υπολογίστηκαν οι συνέπειες για τη δημόσια υγεία του περιορισμού των μέγιστων εκπομπών, όχι μόνο οξυδίων του αζότου, αλλά και μικροσωματιδίων Pax. Άρα, ε, PM, που φάνηκε ότι θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος ο περιορισμός του, των πολύ μεγαλύτερο ο αντίκτυπος του περιορισμού των μικροσωματιδιών από αυτόν του περιορισμού του όζοντος, δηλαδή ε, οξυδίων του αζότου. Οι επιλογές σας λοιπόν στηρίχθηκαν σε μελήματα που γνώμονα είχαν μόνο τη δημόσια υγεία ή και σε τεχνικές δυνατότητες, δηλαδή δυνατότητες να αχνίχνευτούν περισσότερο τα μικροσωματίδια και, το, ή το διοξείδιο του, του αζότου. Και για τον κύριο Μπέ, πέτε μάκι. Οι μέγιστες εκπομπές διοξιδίων ε, οξυδίων του αζότου στα 200 γραμμάρια είχαν κριθεί ως καταλληλότερη επιλογή και αυτό στη μελέτη αντικτύπου 2007 επαναλαμβάνω ή και νωρίτερα ακόμα μπορεί να είναι εφικτό χωρίς να χρειάζεται, χωρίς περαιτέρω κατεργασία SCR δηλαδή. Και ένα όριο των 75 mg το χιλιόμετρο θα κόστιζε 590 ευρώ ανά όχημα για ένα σύστημα after treatment εκ των υστέρων. Και Πρόεδρε, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μπορεί να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως τα 200 μιλιγκράμμα επελέγησαν χωρίς να χρειάζεται το after treatment. Η κυρία Ριβού Νταλόν Μπονφουά. Νταλόν Μπονφουά. Πρόεδρε, ευχαριστώ για τον κανονισμό 715 του 2007 στο άρθρο 13 αναγράφεται ότι τα κράτη-μέλη προσδορίζουν τις παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις. Θεωρείτε ότι επαρκεί αυτό το άρθρο 13 είναι αρκετά ε, σαφές και έχετε ε, καταγράψει τις, τους μηχανισμούς κυρώσεων των κρατών μελών. Από τις επιστολές οχλήσεως που βλέπω να έχετε αποστείλει στα μάλλον δεν διαπιστώσετε καμία τέτοια κύρωση. Επίσης για τεχνικούς ελέγχους, καθώς μιλούμε για ε, νέα οχήματα αλλά και για μεταχειρισμένα που εκπέμπουν περισσότερους ρήπους. Θα υπάρξει ρυθμίση ε, σχετική με το τεχνικό έλεγχο και την τεχνική επαλήθευση αυτών τεχνικών ελέγχων γιατί και εκεί υπάρχουν ε, πιθανότητες απάτης όπως σε παραδείγματι το να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα των ε, εξετάσεων. Σημειώνω δε ότι οι πραγματικέ δοκιμέ, συνθήκε δηλαδή πραγματική οδήγηση, θα πρέπει να υπολογίζονται σε 16 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα, γιατί αυτή είναι η μέση ταχύτητα που μπορεί κανεί να κυκλοφορεί ει Παρισίου. Κύριε Σερτού. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ομολογώ ότι δεν βλέπω διαφορά να είμαι σε μια κανονική συνήθεια επιτροπή και την εξεταστική που έχουμε εδώ. Θα μείνω λοιπόν στο Euro 5, Euro 6 γύρω 5, Euro 6 και θα κάνω την εξής ε, ερώτηση. Είναι ξεκάθαρη στους δύο κανονισμούς η απαγόρευση για τη χρήση μηχανισμών περιορισμού των εκπομπών, με εξαιρέσεις όμως ρητά, που σημαίνουν ε, συγκεκριμένα τη δυνατότητα χρήση μηχανισμών που θα απέτρεπαν την ε, ε, ζημία, πιθανή ζημία στον κινητήρα κτλ. Πάνω σε αυτή την εξαιρεστηρίζονται όλοι οι κατασκευαστέ αυτοκινήτων για να βάλουν αυτού του περιορισμού. Θεωρώ ότι η Επιτροπή τα γνωρίζει αυτά όλα. Πώ λοιπόν μπορεί να αξιολογήσει αυτά τα οχήματα, πού στηρίζονται στην εν λόγω εξαίρεση και τι θεωρεί η Επιτροπή ότι πρέπει να πράξουμε. Τι είναι το πρακτέον, εσεί στη θεματοφύλαξη των συνθηκών, πρόκειται και κανονισμό του 2007. Από το 2007 διαρκώ προβάλλονται επιχειρήματα βάσει αυτών των εξαιρέσεων για να στρεβλώνετε τα αποτελέσματα. Δεν μπορείτε λοιπόν να λέτε ότι δεν υπάρχει μηχανισμός παρέμβασης στην, ε, στα αποτελέσματα. Αντιθέτως, είναι πάγια αυτή η κατάφραση και εσείς ως Επιτροπή τι σκοπεύετε να κάνετε. Και ευχαριστώ. Μεσμάκερ. Δεν Ευχαριστώ. Μία από τις προτεραιότητες μας για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα στη δουλειά, να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν ανεξάρτητη υπήρεξη εφορέας ε, μέτρησης. Είχαμε δοκιμές στηριγμένες σε φορητά συστήματα μέτρηση εκπομπών τα τελευταία χρόνια. σε 1.100 οχήματα, εκ των οποίων το ένα τρίτο ήταν στην Ευρώπη και το άλλο τρίτο και ένα άλλο τρίτο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει λοιπόν κάποια αξιοποίηση από την Επιτροπή αυτών των ανεξάρτητων εκτιμήσεων και υπάρχει περίπτωση αυτές οι ανεξάρτητες δοκιμές που ονομάζονται μάλιστα Emissions Analytics η σχετική εταιρεία. Ε, υπάρχει το να αξιοποιηθεί, γιατί ξέρω ότι πρόκειται να δημοσιεύσει ένα σύστημα βαθμολόγησης για τα οχήματα. Όταν υπάρχουν τέτοια κενά λοιπόν στην Ευρώπη η Επιτροπή σκοπεύει να τα καλύψει αξιοποιώντας αυτούς που κάνουν σωστή δουλειά. Οι συνθήκες επίσης για τις εξαιρέσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρες για να μην γίνονται καταχρήσεις και έχω ερώτηση ως προς την αναγκαιότητα της λεγόμενης λειτουργίας μετάδοσης η οποία δεν διευκολύνει την διαφάνεια. Μπορείτε να μας τα κάνετε πιο λιανά. Ο κύριος Παγνιού, ο κύριος Ζήλ, ε, από τη Πρόεδρε, Μια και σας έχουμε εδώ, όπως λέμε στα γαλλικά, θα σας αξιοποιήσουμε. Λοιπόν, εγώ θα πάω περαιτέρω σε λεπτομέρειες για να στήσω εξηγήσει για να καταλάβω καλύτερα. Πρώτον, πώς οργανώνεται η συμμετοχή των εμπλακωμένων μερών και δι των κατασκευαστών αυτοκινήτων στις τεχνικές συνεδριάσεις της Επιτροπής που, της που ασχολείται με τα οχήματα με κινητήρα, γιατί από αυτά που μαθαίνω Διερωτώ αν οι αρχέ τη χρηστή διοίκηση σε επίπεδο αυτών των επιτροπών έχουν το όντι τσιριθεί. Πρώτον. Δεύτερον, οι κατασκευαστέ και οι οργανισμοί πιστοποίησης πώ οργανώνονται εν ώψη τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων για την του ανταγωνισμό, που πιστεύω ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κάποια πιο χαλαρή αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων. Μην θυμίσουμε τώρα τα επιθέματα από σιλικόνη για το στήθος που ένας γερμανικός οργανισμός πιστοποίησης, ο TÜV, είχε εγκρίνει χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Κύριε Καλέχα, επίσης εσείς αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την ε, επενέσατε για την ε, ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα κτλ. Αλλά, μια και από ό,τι φαίνεται δεν ε, τηρούνται εν γέννη οι προδιαγραφές για, την, ε, για τις εκπομπές των αυτοκινήτων, η άλλη όχθη του Ατλαντικού τι λέει για τις δεσμεύσεις μας σε σχέση με, το, με τις διεθνείς υποχρεώσεις, με την οδηγία ένισε, αφού δεν τηρούνται οι προδιαγραφές του Euro 5 και του Euro 6, ο, η πρόεδρος, έχω ακόμα 7 εγγεγραμμένους ομιλητές και σας καλώ να περιοριστεί το καθένας σε ένα λεπτό. Ο κύριος Σιλικιώτης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσουμε τους διευθυντές για την παρουσία τους εδώ. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχουν και ευθύνε, αλλά υπάρχουν και κενά. Ε, και αποδείχτηκε ότι υπάρχουν κενά στην νομοθεσία. Ε, και που δεν λειτουργούσε αποτελεσματικά με, ευκαιρία, την ευκαιρία να μπορούν οι εταιρείε να ξεφεύγουν του ελέγχου και να κατά την άποψή να έχουν κάλυψη. Δεν ακούσαμε ποια είναι τα κενά αυτή στην νομοθεσία που επιτρέπουν στι εταιρείε να παραβιάζουν του νόμου, που τώρα επιδιώκεται να αλλάξουν για μα έχει ευθύνη και η Κομισιόν και ορισμένε κυβερνήσει. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριο Περτομάκη περισσότερο στι ευθύνε των εταιριών. Στην ερώτηση όμω τη ε, συναδέλφου μου, τη Μέρια, για την Ερευνητική Επιτροπή τη Κομισιόν, δεν απαντήσατε σωστά κύριε Περτομάκη. Η ερευνητική δεν εντόπισε ότι υπάρχει σκάνδαλο. Η Ερευνητική Επιτροπή το 2013 εντόπισε ότι αυτά τα συστήματα τη Volkswagen μπορούν να παραποιήσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Εδώ είναι το ερώτημα. Και γιατί δεν λήφθηκε ε, κανένα μέτρο. Άρα αυτό που ρωτάω και τους τρεις είναι τι είναι εκείνο που θα αλλάξει σήμερα σε σχέση με το τι έγινε ώστε που θα αγγιθεί στο μέλλον αποτελεσματικά το ρόλο τόσο της Κομισιόν όσο και των κρατών μελών. Ιδιαίτερα στα κενά της νομοθεσίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Mr. Κύριο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προσπαθούμε εδώ, σε αυτή την Εξαστική Επιτροπή, να καταλάβουμε τι σφάλματα έγιναν στο παρελθόν, προκειμένου να μην τα επαναλάβουμε στο μέλλον, προκειμένου να καταφέρουμε να επιβάλλουμε τις απαραίτητες κυρώσεις. Και θα ήθελα από αυτού να επιμείνω. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θα είναι ανταγωνιστική, φιλική προς το περιβάλλον όμως παράλληλα. Νομίζω όμως ότι δίνεται εδώ η εντύπωση ότι κάτι παραπάνω πρέπει να κάνουμε. Χρειαζόμαστε ένα άλλο νομοσχετικό σχέδιο. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό θα αποβεί περίπλοκο και χρονοβόρο νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια πρώτη φάση σε έναν τεχνικό εξυγχρονισμό, προκειμένου η αυτοκινητοβιομηχανία μας να αποτελέσει ηγέτη όσον αφορά τις ευφυείς και καθαρείς μεταφορές. Νομίζω ότι διαφαίνεται εδώ πέρα μια ευκαιρία, μια χρυσή ευκαιρία για να κινητοποιήσουμε επιτέλους την Ευρώπη και να μπούμε σε ένα νέο ενάρετο κύκλο όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία. Ο κύριος Σλοτόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητούμε αυτή τη στιγμή τα πρότυπα, τις προδιαγραφές. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και τις διαφορές που υπάρχουν ε, εκτενέστερα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ότι εμείς ασχολούμεθα περισσότερο με, την, ε, με το στάδιο πριν τη διάθεση στην αγορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες το αντίστροφο. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι εδώ πέρα μιλάμε για μια καθερή απάτη. Συσκευές παράκαμψης τοποθετήθηκαν σε οχήματα και ουσιαστικά τροποποιούσαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η ίδια η μηχανή αυτών των οχημάτων με αποτέλεσμα να δίνουν αποτελέσματα πολύ πιο θετικά και πιο αποδεκτά από τα πραγματικά. Έχω λοιπόν μια ερώτηση και δεν ξέρω σε ποιον από τους τρεις σας θα πρέπει να απευθύνω, πάντως είναι η ακόλουθη. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας υφίστανται διατάξεις που θα επέτρεπαν ποτέ την εγκατάσταση τέτοιων συσκευών παράκαμψης ή να το πω διαφορετικά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν διατάξεις νομοθεσία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν δικαιολογία για μια τέτοια δραστηριότητα, που έμεσα θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν, να δικαιολογήσουν μια τέτοια πρακτική. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Παλούτση έχει το λόγο. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Αν κατάλαβα καλά, υπήρχαν όντω πολύ σημαντικέ διαφορέ ανάμεσα στι εργαστηριακέ δοκιμέ και τι δοκιμέ μέτρη σε πραγματικέ συνθήκε οδήγηση και καταβάλλετε προσπάθειε προκειμένου να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα. Ο αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή μα είπε ότι έστειλε και επιστολέ προ τα κράτη-μέλη. Πότε απεστάλησαν αυτέ οι επιστολέ, ποιε ήταν οι απαντήσει που λάβατε από τα κράτη-μέλη επίση. 23 επίσης διαδικασίες επί παραβάση μας είπατε, ή μάλλον επιστολές όχλησης προς ποιους, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ποιος πλήρωσε, επιβλήθηκαν κυρώσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέω κύριος Λόπες. Σαφώ προκύπτει που ακούσαμε ότι κάτι δεν πήγε καλά και τώρα είπαμε θα κατεβάσουμε καινούργια νομοθεσία, καινούριου ε, ελέγχου, καινούργια εποπτεία. Επομένω, όλα αυτά αποδεικνύουν ότι κάτι πήγαινε στραβά. Κάτι πήγαινε στραβά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη. Πού είναι οι συναρμόδιες σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία. Ε, επομένως, εμείς θα πρέπει τώρα να ξεκαθαρίσουμε και να δούμε τι έγινε με, με ε, ποιος φταίει για αυτή την, απάτη και θα πρέπει να πούμε τι, τι, προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε και όσα έγιναν να αποτελέσουν μια ευκαιρία και έτσι τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν για να έχουμε μια αυτοκινητοβιομηχανία πρωτοπόρα. Αυτά γιατί βέβαια αυτή η βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντική για πολλές χώρες και για όλη την ευρωπαϊκή οικονομία. Συγκεκριμένη ερώτηση. Τι μέσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα κρατη και τα θεσμικά όργανα. Τι αρμοδιότητες προβλέπονται για έρευνα και διαπίστωση του κατά πόσο έχουμε χρήση τέτοιων συσκευών. Εδώ υπάρχει κενό, παραθυράκι. Δεν υπάρχουν δηλαδή οι μηχανισμοί που να ε, βοηθούν στον εξωτερικό εντοπιστεί ότι έγινε. Η ε, ε, επόμενη κυρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Διευθυντά, μας είπατε μια κυβερνητική οργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλυψε την απάντηση σε σχέση με τις επίμαχες συσκευέ. Και μας εξηγήσατε και το σύστημα έγκρισης τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς πώς βλέπετε τον ρόλο των μη οργανώσεων όσον αφορά τα αποτελέσματα των δοκιμών, ε, όσον αφορά μέλους της καναγγελίας για απάτη. Φυσικά και εδώ έχουν σαν αρμοδιότητα, είπαμε, για αυτά θεσμικά όργανα και ε, κρατημέλη, αλλά μη κυβερνητικέ οργανώσει τι μπορούν να κάνουν στο μέλλον. Πρόεδρο. Ε, ευχαριστούμε πολύ και τρώχουμε το τελευταίο γύρο. Ε, απαντήσω από τον κύριο Μάκη πρώτα. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε με την ερώτηση του κυρίου Μπελέτα, αξιολόγηση 2007 των συνεπειών, του αντικτύπου και του κόστους ε, για, τις, ε, για την εισαγωγή εκ των υστέρων μηχανισμών. Νομίζω ότι αυτό ισχύει και στη σημερινή μας αξιολόγηση. Άρα, σωστή η παρατήρησή σας. Και βεβαίω θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιες είναι οι τεχνικές λύσεις που θα μπορούσαμε να προτείνουμε, να εισαγάγουμε. Αλλά αυτό ήταν ο τρόπος με τον οποίο έγινε η αξιολόγηση. Κυρώσεις του άρθρου 13. Παρακολουθούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο τις επιβάλλουν τα κράτη-μέλη κανονισμός ε, Euro 5, Euro 6 δεν ήταν τόσο δεσμευτικός, αλλά νομίζω τώρα μετά από αυτό το σκάνδαλο της Volkswagen ε, κοίταμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή να τηρούνται οι απαιτήσει. Για τον Bundestag βεβαίω και παρακολουθούμε τη συζήτηση και τις εξελίξεις. Αντίστοιχα όμως και τις συγκρίσεις μεταξύ ευρωπαϊκού και αμερικανικού δικαίου, γιατί υπάρχουν εξαιρέσει για αυτά τα defeat devices σε ορισμένες περιπτώσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά Νομίζω ότι αυτό είναι και η συζήτηση που διεξάγεται στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Λίγο πολύ. Αυτό έχω να σας απαντήσω προς το παρόν. για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και την ε, διάθεση στο διαδίκτυο των δεδομένων. Βεβαίως και είμαστε, ε, μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τις συνέπειες των μέτρων, να παρακολουθούμε τα σχόλια. Αυτό πρέπει να κάνουν πάντα το δημόσιες αρχές. Και άλλωστε το είδατε, παραπέμψαμε την Γερμανία Παρεπέμφθη η Γερμανία στα δικαστήρια σε περίπτωση ενός ε, συστήματος κινητού κλιματιστικού ε, και μάλιστα αυτό από την ίδια την ε, κατασκευαστική, τον ίδιο το κατασκευαστικό κλάδο. κάτι άλλο. Τα νομοθετικά μέτρα για την, και η παρακολούθηση των ε, εξελίξεων των τεχνολογικών. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Στηρίζομαστε σε αυτό και στο ΚΑΡΣ και στο ΚΑΡΣ 2020 και αργότερα για το 2030. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν και πρέπει να δούμε νομίζω όχι μόνο τα ευφυή αλλά και τα καθαρά οχήματα. Αυτά. Αν δεν έχω ξεχάσει κάτι, θα σταματήσω εδώ. Ναι, θα έλεγα ότι στο αμερικανικό δίκαιο προβλέπεται δυνατότητα χρήση τέτοιων μηχανισμών παράκαμψη ε, σε ορισμένε συγκεκριμένε περιπτώσει όμω. Το βλέπουμε και στον κανονισμό Euro 5-6. Εξαιρετικές περιστάσεις όμως συγκεκριμένες που μπορεί να έχουν να κάνουν με αποτροπή ατυχημάτων, συγκεκριμένους ελέγχους της μηχανής κτλ. Είναι πολύ περιορισμένες αυτές οι χρήσεις της εξαίρεσης. Πάντως εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση σχέση με τη Γερμανία. Είμαστε σε επαφή με τους ε, νομικούς μας συμβούλους και όποτε θέλετε να επανέλθουμε. Ο κύριος Αρτού. Ναι και ευχαριστώ. Λοιπόν που ξαναδεκόπτω. Οι παρεκκλήσει που προβλέπει ο κανονισμός να τι διαβάσει κανεί. δείχνουν ξεκάθαρα ότι κάθε κατασκευαστής και όχι μόνο στη Γερμανία κάθε κατασκευαστής αξιοποιεί καταχράτε αυτής της ε, παρέκκληση που, είναι, που ανέρχεται στο 2007 Ευθύνη λοιπόν δική σας είναι, εάν η εθνική νομοθεσία δεν γραμμίζεται με το δίκαιο, να παρέμβετε. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει, αυτή είναι η συγκεκριμένη ερώτηση. Τι πρέπει να γίνει και γιατί δεν το κάνατε μέχρι τώρα. Απάντηση. Μα ακριβώ αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Ποιε είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες για τι παρεκκλήσει αυτέ που θα επέτρεπαν νομότυπα μια τέτοια παρέκκληση. Γιατί αν δεν είναι νομότυπη παρέκκληση, τότε προφανώς έχουμε να κάνουμε με παραβίαση του δικαίου. Αυτό λοιπόν πρέπει να συμβαίνει. Στοιχεία ακόμα δεν έχουμε στη θέση μας, αλλά τα παρακολουθούμε. Βεβαίως, λέει η Πρόεδρος, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό παρελειμμένος, κατά την εξέταση των θεμάτων αυτών στην Επιτροπή μας στους επόμενους μήνες. Είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε θα μας απασχολήσει. Κύριε Καλέχα. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω τις απαντήσεις του κύριου Περιτομάκη και να απαντήσω και σε ερωτήσεις που απευθύνθηκαν σε μένα. Ο κύριος Μπελέτ πρώτος αναφέρθηκε στη μελέτη αντικτύπου, καθώς επίσης και τις επιπτώσεις στην υγεία από τα οξύδια του αζώτων χρησιμοποίησαμε συγκεκριμένε τεχνολογίες. Μα και τα δύο, και τεχνολογία και τις μελέτες που γίνανε για την υγεία. Θα δείτε ότι τόσο τα οξύδια του αζότου όσο και τα μικροσωματίδια έχουν πολύ δεινέ συνέπειε στην υγεία και προκαλούν προβλήματα βέβαια και στα πλαίσια της, των διζελοκίνητων οχημάτων και γι' αυτό το λόγο στα πλαίσια του RDE, αυτών των νέων δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, θέλουμε προφανώς να μειώσουμε τα επίπεδα και των δύο ουσιών, οξύδια του αζότου και μικροσωματίδια, γιατί έχουν δεινές συνέπειες στην υγεία των πολιτών μας. Απαντώντα σε επόμενη ερώτηση, νομίζω ότι η αναφορά που κάνατε ήταν πάρα πολύ σημαντική σε αυτή την online βάσει δεδομένων όσον αφορά τα PEMS, τα φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών. Η δική μας εσωτερική υπηρεσία έρευνας εξετάζει αυτά τα στοιχεία. Νομίζω όντω ότι θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αυτό το οποίο αναφέρατε. Κύριε Παγνιό, εσείς θέσατε μία ερώτηση για τη συμμετοχή της προσώπων της αυτοκινητοβιομηχανίας στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα της Τεχνικής Επιτροπής για τα οχήματα. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Τεχνική αυτή Επιτροπή συμμετέχει στα πλαίσια της Επιτροπολογίας. Συμμετέχει σε μια άλλη ομάδα διαβούλευσης η αυτοκινητοβιομηχανία, την οποία δημιουργήσαμε το 2011 και ανάλογα τα συμμετοχή τους και στο ΚΑΡΣ 21 και στο ΚΑΡΣ 2020. Ξέρετε ότι ήθιστε να υπάρχουν τέτοιες διαβουλεύσεις με τον κάθε επαγγελματικό κλάδο κάθε φορά. Δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας ή ένας εξωματούχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειώσει τις εκπομπές χωρί να έχει επαφή με του ανθρώπου οι οποίοι εργάζονται στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά δεν αποφασίζει η αυτοκινοβιομηχανία σε καμία περίπτωση και όπω σα είπα, δεν ήταν ικανοποιημένη με τι λύσει οι οποίε υποβλήθηκαν στην αρμόδια τεχνική επιτροπή σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί του και θα σα πούμε και οι ίδιοι ότι δεν ήταν τελικά ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τι λύσει οι οποίε καταλήξαμε. Κύριε Σιλικιώτη, σας θυμάμαι πολύ καλά από τότε που ήσταν ε, υπουργό ε, Βιομηχανίας και είχατε τότε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Μας είπατε τι πρέπει να αλλάξει. Θέσατε ένα πολύ ουσιαστικό ερώτημα. Δύο πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Πρώτον, οι δοκιμές, τα, τα γιατί αυτά τα οποία είχαμε στο παρελθόν δεν λειτουργούσαν. Και δεύτερον, η εποπτεία της αγοράς. Διότι αν έχετε σωστές δοκιμές οι οποίες πραγματικά μετρούν τις πραγματικές εκπομπές σε συνθήκες οδήγησης και από την άλλη έχετε και την απαραίτητη εποπτική αρχή η οποία να λειτουργεί καλά, τότε αποφεύγεται οποιαδήποτε μορφή εξαπάτησης. Και τα δύο όμως αυτή τη στιγμή πρόκειται να γίνουν. Μεταρρύθμιση και του συστήματος έγκρισης τύπου και του συστήματος μέτρησης των εκπομπών. Ο κύριος Τωρίνη μας είπε ότι κάτι παραπάνω πρέπει να γίνει. Μα είπε ότι η νομοθεσία μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, αλλά μπορεί να αποτελέσει αυτή τη στιγμή ευκαιρία για την αυτοκινητοβιομηχανία, αν δηλαδή αρχίσουν και χρησιμοποιούν τη σωστή τεχνολογία. Νομίζω λοιπόν ότι όντω δίνουμε μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή στην αυτοκινητοβιομηχανία να καινοτομήσει και να τι φιλικέ προ τον καταναλωτή λύσει. Ο κύριος Μπλάνκο αλλά και άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο ζήτημα των συσκευών παράκαμψης. Νομίζω ότι πρέπει να σας δώσω εδώ μια ξεκάθαρη απάντηση. Αυτές οι συσκευές εξαπάντησης, οι συσκευές παράκαμψης απαγορεύονται από το 2007 και μετά στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου. Και μάλιστα από το 2007 και μετά οποιοδήποτε χρησιμοποιεί τέτοιες συσκευές ουσιαστικά παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο και μπορεί να το επιβληθούν και συγκεκριμένε κυρώσει. Ποιο επιβάλλει τι κυρώσει αυτέ, τα κράτη-μέλη. Γιατί τα κράτη-μέλη, γιατί αυτά κάνουν την έγκριση τύπου. Τα κράτη-μέλη λοιπόν αυτά που πρέπει να ελέγξουν ότι όντω τα οχήματα δεν φέρουν συσκευέ παράκαμψη, συσκευέ εξαπάτηση. Α μην υπάρχει καμία παρανόηση επ' αυτού. Αν εξαπατά ένας κατασκευαστής οχημάτων, τότε επ' αυτού πρέπει να επιβληθούν κυρώσει γιατί αυτές οι συσκευές, το παραλαμβάνω, απαγορεύονται ρητά στα πλαίσια του ουσιακού δικαίου και αυτό έχουμε επαναλάβει ρητός πάρα πολλές φορές. Ο κύριος Μπλάνκο έθεσε ένα ερώτημα. Ποιος έφταιγε τα κρατημέλη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα κοιτάξτε, εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια περίπτωση, ξεκάθαρη περίπτωση απάτης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν κάποιος κινείται παράνομα τελικά, τότε αυτός φταίει. Τι πρέπει εμεί να κάνουμε, να εξασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Και πώ θα γίνει αυτό, βελτιώνοντα την κοινοτική νομοθεσία, βελτιώνοντα τα τεστ που χρησιμοποιούμε, καθώ επίση και του μηχανισμού εποπτεία τη αγορά. Αν δεν καταφέρουμε να διορθώσουμε τα πράγματα και στου τρει αυτού τομεί, τότε δεν πρόκειται να διορθώσουμε τίποτα. Οπότε απεστάλησαν οι επιστολέ ήδη τον Ιούλιο του 2012 ο έγραφε προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη εποπτεία όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία. Εκεί ότι θα πρέπει να αλλάξει και ο μηχανισμός εποπτείας της αγοράς για τα οχήματα, πρόταση η οποία μπλοκαρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 23 επιστολές στείλαμε όσον αφορά τις ε, κυρώσει και προχωρήσαμε σε κάποιες πιλωτικές διαδικασίες όσον αφορά τις παραβάσεις. Κυρία Σαλτεμόσε, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν μπορούμε να εργαστούμε χωρίς αυτές. Αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα του όλου συστήματος, μας βοηθούν πραγματικά να θέτουμε τα πράγματα στο σωστό τους πλαίσιο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και να συμμετέχουν και πραγματικά να καταγγέλουν τα κακό κείμενα. Εγώ πριν από οποιοδήποτε Συμβούλιο Περιβάλλοντος συζητώ με προσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων, έχουμε τακτικό διάλογο μαζί τους, αλλά και σε προηγούμενα πόστα που είχα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσα ότι πάντα ήταν πολύ σημαντικό να ακούμε τους πάντες. Συλλόγους καταναλωτών, βιομηχανία, επαγγελματικό κλάδο, αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Διαφορετικά δεν καταφέρνουμε τίποτα να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει Κύριε θέλετε να ξαναπάρετε το λόγο ο κύριος Μέτσκερ, με συγχωρείτε, όχι, δεν επιθυμώ να ξαναπάρω το λόγο. Θα μπορούσαμε να θέσουμε και περαιτέρω ερωτήσεις, αλλά όπως σας είπα, πρόκειται για την πρώτη επαφή που έχουμε προσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι θα επαναληφθούν και στις επόμενες συνεδριάσεις μας όλες αυτές οι ερωτήσεις, θα προκύψουν πάλι με τον ένα τον άλλο τρόπο, αν εκκρεμούν αυτή τη στιγμή οι περαιτέρω ερωτήσει που θα θέλετε να θέσετε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορείτε να τι θέσετε γραπτώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει και όλοι θα έχουν πρόσβαση και σε ερωτήσει και σε απαντήσει σε συνθήκε απόλυτη διαφάνεια. Όπως σας είπα θα απαντηθούν ε, περαιτέρω τα ζητήματα αυτά και σε επόμενες συνεδράσεις. Θα περάσουμε τώρα και στο πρόγραμμα εργασίας μας. Καταρχάς όμως να ευχαριστήσω τους τρεις εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαθέσιμότητά τους, για τον ιδιαίτερα ανοιχτό τρόπο με τον οποίο απάντησαν και το γεγονό ότι πολλέ φορέ δεν έχουν οι ίδιοι βέβαια τι απαντήσει, Για τι απαντήσει σε κάποια ερωτήματα έπρεπε να δώσουν ή τα κράτη-μέλη ή εκπρόσωποι τη αυτοκινητοβιομηχανία. Για άλλη μια φορά όμως ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα και πιστεύω θα σας ξαναδώ πολύ σύντομα μέσα στους επόμενους μήνες. vice uh, Οι αντιπρόεδροι μπορεί να έρθουν ε, εδώ στο Προεδρείο γιατί αισθάνομαι λίγο μόνοι. Okay, colleagues. Uh, let's move on. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε, ας περάσουμε στο τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό σημείο της ημερήσιας διάταξης, μελλοντικό σχέδιο εργασίας. Θα γνωρίζετε ενδεχομένω από τους συντονιστές σας ότι κάναμε ήδη κάποιες συναντήσεις, μία μάλιστα σήμερα το πρωί, προκειμένου να θεσπίσουμε το πρόγραμμα εργασίας μας και τις μεθόδους εργασίας μας για το υπόλοιπο του έτους. Και ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το εγχείρημα δεν είναι καθόλου εύκολο. Ζητήσαμε λοιπόν από όλες τις πολιτικές ομάδες να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι τις 22 Μαρτίου για να δούμε ποιους εμπειρογνώμονες θα καλέσουμε στις ακροάσεις μας και είπαμε ότι θα πρέπει πρωταρχικά να εστιαστούμε στο πρώτο ίμιση του 2016. Βρισκόμαστε λοιπόν εν μέσω διαδικασίας αυτής. Πρέπει να σας πω καταρχάς ότι στην επόμενη συνεδρίαση που είναι στις 19 Απριλίου Έχουμε ήδη καθορίσει την διεξαγωγή της πρώτης δημόσιας ακρόασης με το JRC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές μας, οι οποίοι μπορούν να μας πούνε πώς έχουν τα πράγματα, που έχουν εντοπιστεί προβλήματα Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις παρατηρήσεις που υποβάλλατε για το σχέδιο εργασίας μας. Και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα έχουμε ακόμα μια συνάντηση των συντονιστών προκειμένου να καθορίσουμε τη μεθοδολογία μας για τις ακροάσεις που θα γίνουν το πρώτο ήμιση του έτους. Πρώτα ο κύριο Ζάλμπα και μετά ο κύριο Γκερμπράντι. Ευχαριστώ. Κύριο Χερμπράντη, κύριε Παφενόμενο, πρέπει να σα εξηγήσουμε την πρότασή μα για τη μεθοδολογία των αμέσω επομένων ε, μηνών. Ε, θα είναι στενή η συνεργασία μα και θα συνεργαστούμε μεταξύ μα και με του ηγητές. Όλοι γνωρίζουμε και έχουμε διαβάσει στον τύπο το ποια θα είναι τα προβλήματα, οι προκλήσει των μέσων επομένων μηνών. Υπάρχουν προσδοκίε για το έργο τη Επιτροπή μα και νομίζω επομένως ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε και να σταθούμε στο ύψος αυτών των προσδοχιών. Είναι πολύ σημαντικός ο κλάδος του αυτοκινήτου για το μέλλον της ε, Ένωσης και επίσης για το μέλλον ε, όλων αυτών των εργαζομένων. Επίσης γνωρίζουμε για το ότι αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να ε, επενδύσει σε έρευνα. Κρίση και ευκαιρία. Καμία αμφιβολία δεν διατηρώ. Αλλά επίσης και ότι αυτή η κρίση δεν θα πρέπει να οδηγήσει ε, στο να απειληθεί και μία θέση απασχόληση στην Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να συζητήσουμε τώρα ποιο θα είναι το φύλλο πορεία, ο χάρτη πορεία για του επόμενου μήνε. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Χερμπράντη, με την ε, πρόεδρο και με τους ε, εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Νομίζω ότι τα έχουμε συμφωνήσει και είναι ισορροπημένο το αποτέλεσμα. Άρα τον Ιούνιο θα κάνουμε το συμπίλημα όλων των πληροφοριών και έτσι θα καταλήξουμε σε κάποια γνωμοδότηση. Οπότε και θα είναι όσο γίνεται πιο στεγανό το έργο μας. Έχουμε τρεις άξονες τώρα. Πρώτα-πρώτα θα συμβουλευτούμε κάποιους ειδικού για τεχνολογία που αφορά τους κινητήρες των αυτοκινήτων. Δεύτερος άξονας θα είναι κάποιες ακροάσεις με ειδικού όσον αφορά τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες. Τρίτος άξονας ε, των ακροάσεων θα είναι ειδική για τη μόλυνση και ρήπανση της ατμόσφαιρας. Όλοι αυτοί οι ειδικοί πρόκειται να μας εκθέσουν τους απόψεις, όμως κατά το δεύτερο ημιση του έτους θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με επιτρόπους. Και θα επεξεργαστούμε κάποιες ερωτήσεις προς κρατημέλη. Και θα τα συζητήσουμε κατά τις αποστολές που θα κάνουμε προς τα κρατημέλη. Τέλος εγώ και τώρα τη σκητάλη που παίρνει ο κύριος Χερμπράντι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ Παύλο Σάλβα. Ξεκινώ λοιπόν πρώτον για να αποφύγουμε τις μείζονε απογοητεύσεις. Τώρα έρθει η ώρα για την ενδιάμεση έκθεση. Ενημερώνω τους πάντες ότι δεν θα έχει πολιτική χρειά αυτή η ενδιάμεση η έκθεση. Είναι υποχρεωτικό λόγω του ιστορικού μας να εκδοθεί ενδιάμεση έκθεση, αλλά έχουμε αποφασίσει να μην την καταστήσουμε, να μην ακολουθήσουμε μια υψηλών τόνων πολιτική. Αυτό, για να μην μπερδευόμαστε και απογοητευόμαστε. Δεύτερον, η σειρά με την οποία οργανώνουμε τις ακροάσεις και τα ονόματα των προσκεκλημένων φυσικά έχουν τεράστια σημασία Γι' αυτό και αποφασίσαμε να ζητήσουμε από τους συντονιστές και το ακολουθούν οι συντονιστές και το ανέφερε ήδη συνάδελφος. Να ξεκινούμε με τους τεχνικούς λεγόμενους εμπειρογνώμονες για την τεχνολογία των κινητήρων, για τις εκπομπές σε, και τις μετρήσεις τους σε πραγματικές συνθήκες. Με αυτό ξεκινάμε λοιπόν. Περνάμε στη συνέχεια στα πιο πολιτικού χαρακτήρα ζητήματα, στα οποία εγώ εντάσσω και την κοινωνία των πολιτών. Και έτσι θα στραφούμε προς την κοινωνία των πολιτών για πρώτη φορά. Με εκπροσώπους από τις ΗΠΑ, υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας. Για να δούμε και τι νομοθεσία ισχύει εκεί και τι Διαφορές υπάρχουν. Και θα κοιτάξουμε και όχι μόνο την Επιτροπή και τους ειδικού της, αλλά και άλλους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και οργανώσεις πολιτών. Μετά έχουμε μια ομάδα που θα εκπροσωπήσει τον, τον κλάδο της βιομηχανίας και μετά, φθινόπορο πια στα τέλη, θα έχουμε τους επιτρόπους. Αυτό είναι μια όχι μόνο χρονολογική σειρά, αλλά και η έκφραση μιας στρατηγικής σκέψης πίσω από την ε, τάξη αυτή, τη σειρά αυτή. Και χαιρόμαστε που έγινε δεκτή αυτή. Ναι, αν μου επιτρέπετε θέλω και εγώ να ενημερώσω ότι κάθε χρόνο οργανωνόμαστε ως Επιτροπή για να καταθέσουμε ερωτήσεις με βάση βέβαια τις προτάσεις των πολιτικών ομάδων να έχουμε δέκα ή περισσότερες ερωτήσεις που θα κατατεθούν προκαταβολικά ενώ κάθε συνεδριάσεως και θα λάβουν γραπτές απαντήσεις ώστε να είμαστε έτοιμοι και να αξιοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά το χρόνο μας. Αυτό για να ξέρετε δηλαδή ότι θα σας ε, Προτείνουμε ερωτήσει εν ώψη της προετοιμασίας των συνεδριάσεων. Δεύτερον, είναι σημαντικό επίση να έχουμε τιμονό ερωτηματολόγιο, απευθυνόμενο στα κράτη-μέλη αυτή τη φορά, για τους τύπους των εγκρίσεων, για την εποπτεία της αγοράς κλπ. Κοιτάμε λίγο πώς θα το χειριστούμε, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, αλλά πάντως βασικό είναι πριν έρθουν στην Επιτροπή για μια ακρόαση οι εκπρόσωποι και όπως είπα είναι περιορισμένος ο χρόνος μέσα στις εκροάσεις μας και είναι απαραίτητο να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, να ξέρουμε τι είδου απαντήσεις δίνονται σε πρώτη δόση στις ερωτήσεις μας για να μπορούμε να ε, υποβάλουμε συμπληρωματικές. Αυτά λοιπόν προς την προετοιμασία. Πολιτικές ομάδες, παρακαλώ. Κύριε Σκίσεκε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Υποστηρίζουμε πλήρως ε, τις επιλογές των δύο συγκητών μας, βεβαίως καταρχήν. Είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Ε, μια ε, θεμελιώδη μόνο παρατήρηση θα ήθελα να διατυπώσω ότι έχουμε μια σαφή εντολή και δεν πρέπει από αυτή να παρεκκλίνουμε. Εμεί ω ΕΛΚ θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να αποδηθεί σε ένα κυνήγη μαγισσών η Επιτροπή μας. συγκεκριμένα περιστατικά εξετάζει, συγκεκριμένες πράξεις εκμερών ατόμων και με αυτό το δεδομένο προχωρούμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε δηλαδή μια πολιτική αμάυρωση ενός ολόκληρου κλάδου ε, ή να καταγγείλουμε όλη τη βιομηχανική παραγωγή της Ευρώπης. Τελευταία ανάλυση πρόκειται για πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Πρόκειται για μια ε, συγκεκριμένη περίπτωση την οποία θέλουμε πρακτικά να αντιμετωπίσουμε. Επίσης δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα περιοδεύοντα θεία σου αυτή η Επιτροπή, εάν χρειάζεται να επισκεφθούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν χρειάζεται να μιλήσουμε με τους Αμερικανούς, ε, δεν χρειάζεται να πάει η μισή Επιτροπή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας τους καλέσουμε δύο-τρεις ανθρώπους να έρθουν εδώ να μας μιλήσουμε. Αυτά επικοδομητικά από πλευράς του ΕΛΚ. Βεβαίως, βεβαίως και ευχαριστώ και επιπλέον Εάν έρθουν εδώ οι ειδικοί από τι ΗΠΑ, συμπληρώνω, θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν ερωτήσεις. Αυτό ενισχύει και τη διαφάνεια. Κύριε Ντάνς. Δεν έχω πολλά να προσθέσω βεβαίως προς συμφέρον όλων των ομάδων. Να επιτελέσω σωστά το έργο της αυτή η Επιτροπή δηλαδή στο τέλος της να υπάρχει, να έχει ανακτηθεί η εμπιστοσύνη, η αξιοπιστία των κατασκευαστών έναντι του καταναλωτή. Νομίζω ότι και στους συντονιστέ υπόθηκαν πολλά και επικοδομητικά εν ώψη της προετοιμασίας της ε, έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής μας. Βασική αρχή είναι ότι συλλέγουμε δεδομένα και μαρτυρίες και στοιχεία στην πρώτη φάση για να τα έχουμε όλα στη θέση μας όταν έρθει η ώρα να τα ε, προβάλλουμε σε εκείνους που βρίσκονται στην κατάλληλη θέση για να μας δώσουν απαντήσεις και να καταλάβουμε και τι είδους απαντήσεις μας δίνουν. Αναφέρθηκε ήδη παρατήρηση σχετικά με τις αποστολές. Ναι, Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε στο δυνατόν λιγότερο να μετακινούμαστε εμείς. Αλλά μπορεί να πάμε στο Λουξεμβούργο, Φερρυπίνη. συναρπαστικό και αυτό το ταξίδι. Αλλά και την Ιταλία θα πρέπει να επισκεφθούμε. Και νομίζω πρέπει να ενσωματώσουμε την αρχή αυτή, να δεχθούμε την αρχή αυτή, να προσκαλούμε δηλαδή εδώ τους ε, Αμερικανούς που θα θέλησουμε να ακούσουμε και όχι να χρειαστεί εμείς να πάμε εκεί. Πάντως βασική αρχή θα πρέπει να είναι να μην αφήσουμε την ανάγκη να παραχθεί μια έκθεση να επηρεάσει την τεχνική αρτιότητα της δουλειάς που θα κάνουμε εδώ. Και πρέπει να ε, μεριμνήσουμε να λάβουμε επακριβείς απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Πρέπει να έχουμε επαρκή χρόνο και για τις ε, παρουσιάσεις για τις απαντήσεις τους, αλλά και για ενδεχόμενες συμπληρωματικές ερωτήσεις, ώστε να επαληθεύουμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να κλείνουμε τουλάχιστον δύο μέρες συνεδρίασης για την Επιτροπή, με βάση και τις ερωτήσεις βεβαίως που θα έχουμε προκαταβολικά καταθέσει, γιατί έτσι μπορεί κανείς να κοιτάξει λεπτομέρειες με βάση τις γραπτές απαντήσεις, με συγκεκριμένους μάρτυρες, που είναι απαραίτητη βεβαίω εάν θέλουμε να έχουμε και συγκεκριμένε απαντήσει. Ο κύριος Ροσφόρο επιθυμεί να πάρει το λόγο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ξεκινάμε πολύ καλά τις εργασίες μας. Να συγχαρώ εκ των προτέρων τους δύο εισηγητές, όχι προφανώς για την τελική τους έκθεση, αλλά για τη μέθοδο την οποία προετοίμασαν από κοινού. Οι συνάδελφοι έχουν απόλυτο δίκιο όταν λένε ότι θα πρέπει να μην χάσουμε τους βασικούς μας στόχους από την προσοχή μας. Πρέπει να δούμε πραγματικά εδώ πέρα πού θέλουμε να κινηθεί αυτή η Επιτροπή. Πρέπει να δημιουργήσουμε πρότυπα και τα πρότυπα αυτά έχουν να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον, με το κοινό καλό. Στη συνέχεια τα πρότυπα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν. Αυτό μας απασχολεί κυρίως, πώς θα εφαρμόσουμε σωστά αυτά τα πρότυπα. Ξέρετε ότι όταν τα πρότυπα χρησιμοποιούνται σωστά μπορούν να αποτελέσουν και εμπορικό επιχείρημα για τους ίδιους κατασκευαστές. Προωθούν προϊόντα πλέον τα οποία είναι πιο ποιοτικά. Νομίζω λοιπόν ότι οι ψηφοφόροι μας, οι οποίοι είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες και είναι και καταναλωτές, επιθυμούν να δούνε κάτι τέτοιο. Τα, όταν δημιουργούμε πρότυπα, τα πρότυπα αυτά πραγματικά να περνούν έπειτα και στα προϊόντα και εμπροκειμένου στα οχήματα. Και πρέπει νομίζω να έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά η οποία θα είναι ισότιμη. Τι σημαίνει αυτό. Όλοι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι που θα πρέπει να χρησιμοποιούν συσκευές απαγορευμένες καταλαβαίνετε ότι αυτό θα, είναι αθέμητο και θα πρέπει να αποκλειστούν από την αγορά. Επίσης, σε ορισμένα κράτη-μέλη πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό και θα πρέπει να δούμε τι δουλειά έχουν κάνει. Δύο χώρε, το Βέλγιο και η Γαλλία, έχουν δημιουργήσει ειδικέ επιτροπέ για το ζήτημα αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε σε επαφή με τι κοινοβουλευτικέ αυτέ επιτροπέ στο εθνικό επίπεδο. Δεν ξέρω πώ θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να βλέπουμε την ίδια καρικατούρα που είδαμε πριν από λίγο, δηλαδή επικαλύψεις ανάμεσα στο εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο, η έλλειψη συντονισμού. Και πέρα από τις δύο αυτές χώρες υπάρχουν πέντε ακόμα χώρες στις οποίες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για το ζήτημα που μας απασχολεί εδώ. Ουσιαστικά για το σκάνδαλο αυτό, ας το πούμε με το όνομά του. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι δεν εργαζόμαστε εδώ πέρα απομονωμένοι, ξεχωριστά από όλου του άλλου, αλλά θα πρέπει από κοινού να δούμε τι κάνουν και εθνικοί βουλευτέ σε ορισμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ντελή, έχει το λόγο. Όχι, Η κυρία Κιλιόνεν πρώτη, με συγχωρείτε. Μην ανησυχείτε, <laughs> είμαι και τόσο ευαίσθητη. Όχι, όχι, όχι, κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό για μένα να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Θα μιλήσω φιλανδικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θεωρώ ότι έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Καταλαβαίνετε ότι οι προσδοκίες βέβαια από την Επιτροπή μας είναι τεράστιες. Οι φορολογούμενοι Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές περιμένουν από εμά να εξασφαλίσουμε ότι όντως οι κανόνες θα τηρούνται. Και πραγματικά ως φορολογούμενοι ή ως καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τι πληρώνουν και γιατί. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί πάρα πολλούς Ευρωπαίους εργαζόμενους. Και για αυτούς λοιπόν προ το δικό του το όφελο πρέπει να εργαστούμε, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να καταφέρουν να διατηρήσουν τη θέση απασχόλησή του στον τομέα τη μηχανία. και μέσω τη καινοτομία των νέων τεχνολογικών εφαρμογών. Ελπίζω θα καταλήξουμε τελικά σε αυτοκίνητα, σε οχήματα τα οποία θα είναι πιο φιλικά προ το περιβάλλον στο μέλλον. Η δική μου πολιτική ομάδα είναι ικανοποιημένη από το προτινόμενο σχέδιο εργασία και από τι προτινόμενε δημόσιες ακροάσεις και ελπίζω ότι μέσω του προγράμματος αυτού θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε σε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει στα πλαίσια της Εξαστικής μας Επιτροπής και ότι θα πετύχουμε τους στόχους αυτούς στα πλαίσια μιας επικοδομητικής θετικής συνεργασίας χωρίς να αναλωνόμαστε σε αψιμαχίες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν πολίτες, εργαζόμενοι, εργοδότες περιμένουν θετικά αποτελέσματα από το δικό μας το έργο. Η κυρία Ρέντα έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάει ο χρόνος, πιέζει ο χρόνος, πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Και το πιο σημαντικό στα πλαίσια της δουλειάς μας είναι να καταφέρουμε να έχουμε όλα τα απαραίτητα αποδεκτικά στοιχεία αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κάνουμε ερωτήσεις προς αυτούς τους οποίους πρέπει τελικά εμείς να ερευνήσουμε περισσότερο, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία, τα απαραίτητα έγγραφα. Συμφωνώ λοιπόν με τους συζητητές ότι θα πρέπει ερωτήσεις να θέσουμε στους υπευθύνους κάποια στιγμή στα πλαίσια της εργασίας μας, αλλά θα πρέπει να εξερθολογήσουμε και τη διαδικασία απέτηση εγγράφων. Αν όλα περνούν μέσω της γραμματείας, τότε αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, να χρησιμοποιούμε όλη τη μέθοδο αυτή και να μην έχουμε καθυστερήσει όσον αφορά την υποβολή των εγγράφων. Όσον αφορά τώρα τις επισκέψεις, αντιπροσωπείες, Χαίρομαι πάρα πολύ που η EPA και όχι το ΕΛΚΟ, όπω είπε η ομιλήτρια, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και νομίζω το έχουμε δει και από άλλε επιτροπέ ότι είναι πολύ σημαντικό μια εξεταστική επιτροπή να μπορεί να κάνει και διερευνητικέ αποστολέ. Προφανώ λοιπόν θα πρέπει να πάμε σε κάποιε χώρε, αλλά βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε σε αυτέ τι αποστολέ αν δεν το επιθυμείτε, αν δεν το βρίσκετε χρήσιμο. Τώρα, όσον αφορά αυτό το call of evidence που είπαμε, την ε, συγκέντρωση αποδεκτικών στοιχείων. Να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο αυτή, αλλά να υπάρχει και το απαραίτητο επίπεδο εμπιστοσύνη. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στα πλαίσια της αυτοκινητοβιομηχανίας οι οποίοι δεσμεύονται από ε, συμφωνίες ε, επί απορρίτων δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει απαραίτητη εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών και ημών, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η ανταλλαγή αυτή εγγράφων, αν όχι μέσω της ηλεκτρονικής οδού, τότε με, τον κλασικό τρόπο, με την αποστολή δηλαδή συγκεκριμένων εγγράφων σε εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, σωστή τι ερώτηση, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ανωνυμία. Δεν είναι εύκολο πάντως. Θα το προσπαθήσουμε, άλλωστε έχουμε να που να υποβάλουμε στην νομική υπηρεσία. Θα το, θα το παλέψουμε. Είναι μία από τις πολλές δυσκολίες που έχουμε, αλλά θα το κοιτάξουμε. Εγώ. Ναι, τι θα γίνει με αυτό το θέμα του κατά πόσον θα μπορέσουμε να καλέσουμε τόσες ακροάσεις τους βουλευτές, τους ε, εθνικούς. Άλλωστε και στα Εθνικά Κοινοβούλια γίνονται τέτοιες ε, εξεταστικές επιτροπές, οπότε θα μπορούσαμε να συντονιστούμε και σε κάποιο από το πρώτο το δεύτερο ήμιση της χρονιάς θα είναι χρήσιμο το να συντονιστούμε κατά αυτόν τον τρόπο εκεί όπου γίνεται τέτοιο έργο από τους εθνικούς βουλευτάς. Δεν έχω εγώ παρατηρήσεις ε, για την μεθοδολογία, τη διαδικασία. Εγώ στην ΙΜΚΟ εργάζομαι και έχω αναλάβει την νομοθεσία τη σχετική με τα οχήματα και την έγκριση τύπου Οπότε θα ξεκινήσουμε ε, αυτή την διαδρομή μέσα από το Στρασβούργο στην ΙΜΚΟ. Πολύ σημαντικά τόσο σήμερα ακούσαμε ότι πολλές από τις λύσεις έχουν προταθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς τα συντάσματά μας, οι προτάσεις μας θα ληφθούν υπόψη. Άρα ίσως θα πρέπει η ΙΜΚΟ να αναβάλει προς το παρόν τη δουλειά για την έγκριση τύπου. Δεν ξέρω αν νομίζω ότι αυτό είναι ρεαλιστικό και έτσι να μην ε, πάει χαμένη δουλειά που κάνουμε εδώ. Δηλαδή, αυτά στο οποίο θα καταλήξουμε να μπουν στην καινούργια πρόταση. Αυτό θα το συζητήσουμε τους δύο σύγκριτες, λέει ο Πρόεδρος. Και με την ε, διάσημη CCC, την Επιτροπή δηλαδή, των Πρόεδρων των Επιτροπών, τη διάσκεψη των, Επιτροπών τέλο πάντων. Ε, βέβαια, μην προχωρήσει ακριβώς αυτή η νομοθετική πρόταση, ενώ εμείς ε, ερευνούμε τα σχετικά προβλήματα. Θα το λάβουμε υπόψη αυτό που είπατε. Άλλος. Θέλει το λόγο πριν ευθερολογήσουν οι συγκητές. Όχι. Επομένως. Κύριος Θάλμπα γαρε Το λόγο εκεί. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, οι οποίοι υπέβαλαν ερωτήσεις για το θέμα. Πολύ σημαντικό επικοδομητικά να συνεργαστούμε όλες οι πολιτικές ομάδες. Βεβαίως θα έρθουν υπόψη όλα όσα ακούσαμε απόψε. Ο κύριος Χερμπράντι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Απλώς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Και η πρόταση το να καλέσουμε εθνικού βουλευτές ναι, στέγη γιατί γίνονται εξεταστικές επιτροπές και σε μια σειρά εθνικών κοινοβουλίων τώρα. Οπότε ναι και εμείς έχουμε κατά νου να καλύψουμε, να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα εκείνων των επιτροπών. Όπως είπε και ο Πρόεδρος όμως, θα πρέπει να κάνουμε μια συνάντηση με κάποια εθνικά κοινοβούλια. Αλλά πάντως ευχαριστούμε για την πρόταση, του Πρόεδρος όλες που θα σταλθούν υπόψη συνάδελφοι γιατί πολλά θα πρέπει να αποφασιστούν. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε συνεδρίαση και θα γίνει αυτό, αλλά και πάρα πέρα. Και τη μέθα επόμενη και στο μέλλον. 19 Απριλίου είναι η επόμενη συνεδρίαση. 19 Απριλίου. Εκεί θα έχουμε μια αυθεντική ακρόαση, καταθέσεις, εμάρτυρες. Οπότε και έτσι θα καθιερωθούν κάποιοι κανόνε που θα ισχύσουν και στο μέλλον. Παρακαλώ όλοι να έρθετε εδώ διαβασμένοι, να έχετε διαβάσει τις, ε, ε, κατάγραφα των ερωτήσεων που θα βγουν από του ε, Οπότε παρακαλώ όλοι, οι πολιτικέ ομάδε και συντονιστέ, και όλοι να οργανωθούμε. Να, να προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα. Είδατε, σήμερα ήταν πολύ καλή η συζήτηση και ανοιχτή. Αλλά, αλλά, είχαμε πολλές επικαλύψεις ερωτήσεις, αλλά ούτε απαντήθηκαν και όλες οι ερωτήσεις. Γιατί εκείνη η, η κατάθεση, η, συγγνώμη, ακρόαση για, του, για τους μάρτυρες θα πρέπει να πάει όσο γίνεται πιο βαθιά, θα πρέπει να ε, συλλέξουμε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία. Παρακαλώ, προετοιμαστείτε όσο γίνεται καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοδομητική συνάντηση. Θα τα πούμε στο Στρασβούργο. Στου διαδρόμου, αλλά και στι 19 Τετάρτου για την επόμενη συνεδρία. Σε ευχαριστώ. Ξέχασα τίποτα.